Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε κατευθείαν στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ε, θα ξεκινήσουμε λίγο καθυστερημένα την απογευματινή μας συνεδρία ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Γενικός Γραμματέας της IPU, κύριος Τζόνσον, ε, θα είναι κοντά μας και σήμερα το απόγευμα για να εξετάσουμε το θέμα μας που αναγράφεται στο πρόγραμμα και θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία, με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που είναι ε, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και είναι, ήταν, υπήρξε επίσης και δήμαρχος της Αθήνας. Ε, δεξιά μου είναι ο κύριος Μορέιρα, πρόεδρος ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συναδελφός μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ο κύριος Μασελ Ποπόσκι από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. και ο Γιάνν Βάουτερς, ε, καθηγητής στην έδρα Μονέ για το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Οργανισμούς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπακογιάννη. Θα κάνει μια πρώτη εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω μέρος σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Ακόμα και μετά το γεύμα εντυπωσιάζομαι από την παρουσία σας εδώ. Ε, Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ε, γεύμα και ο κύριος Μπρόκ έκανε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία. Είχα προετοιμάσει και εγώ μια ομιλία, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιες απαντήσεις ε, στις οποίες, τις οποίες έθεσε ο κύριος Μπρόκ. Όλοι μας γνωρίζετε, Πρόεδρε, ότι βιώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική κρίση, μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή κρίση. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται επίσης και μια κρίση νομιμοποίησης. Και τίθεται ένα θέμα εδώ, τι μπορεί ένα μέλος του Κοινοβουλίου όπως εγώ να κάνει για να δώσει απαντήσεις στα ερωτηματικά τα οποία θέτουν οι πολίτες. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα, στα οποία δεν ξέρω ότι έχουμε, δεν, δεν βλέπουμε απάντηση, είναι ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνεται σαν να είναι πολύ μακριά από το λαό. Και θα πάρω παράδειγμα τη χώρα μου. Φυσικά η χώρα μου περνάει από μια πάρα πολύ σκληρή κρίση όπως ξέρετε. Βρισκόμαστε στο πέμπτο έτος της ύφεση. Έχουμε 60% άνεργους νέους. Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Ο κόσμος έχει χάσει το 35% του εισοδήματός του. Γενικά ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Φυσικά υπήρξε η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσήλθε, μας βοήθησε και μας υποστήριξε. Όμως τελικά υπήρξε ένα κενό. Υπήρξε ένα κενό, ένα ρήγμα ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες έβλεπαν την κατάσταση και στον τρόπο με τον οποίο ε, τα υπόλοιπα κοινοβούλια ε, της Ευρώπης έβλεπαν ε, την κατάσταση στην Ελλάδα. Και δεν αναφέρουμε μόνο στα μέσα ενημέρωσης όπου η Ελλάδα υπέστη επιθέσεις σαν το μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής οικογένειας, οι τεμπέληδες που κάνουν ηλιοθεραπεία και οι άλλοι πληρώνουν τα σπασμένα κτλ. Σε θέματα πιο σοβαρά υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε εμείς τα πράγματα και οι εταίροι μας. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν έτσι ώστε να κατανοούμε καλύτερα οι μεν τους δε. Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε οι λαοί και οι κοινωνίες μας να κατανοήσουν και να γνωρίζουν την πραγματικότητα στις διάφορες χώρες μας. Κατά τη γνώμη μου εδώ χρειάζονται τα κοινοβούλια των κρατών μελών περισσότερο από ό,τι αυτό γίνεται σήμερα. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται οι ευρωβουλευτές, άμεσα εκλεγμένοι και ότι φέρνουν στην επικαιρότητα πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις χώρες τους, πολύ περίπλοκα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τα κοινοβούλια των κρατών μελών αισθάνονται ότι αγνοούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και θα πρέπει να πω εδώ ότι το κοινοβούλιο μας, η Βουλή των Ελλήνων, τα τελευταία χρόνια ένιωσε σαν να είναι απλά μία μηχανή ψηφοφορίας. Απλά μας ζητούσαν να ψηφίζουμε μία νομοθεσία η οποία μας επευλήθη. Μία νομοθεσία η οποία κάθε φορά μας επιβάλλεται από τους δανειστές. Δεν ζητήθηκε η γνώμη μας. Δεν ε, λήφθη υπόψη η γνώμη μας. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν η Βουλή των Ελλήνων είχε πραγματικά ληφθεί υπόψη, οι απόψεις της, πολλά από τα λάθη τα οποία έγιναν στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και στα πλαίσια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Τρόικα, θα είχαν αποφευθεί κάποια από αυτά τα λάθη. Για να μην μακρηγορώ, να σας πω ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να γίνουν πρωτοπόροι Πώς θα το κάνουν αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να εμπλακούν πολύ περισσότερο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, γιατί κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σήμερα. Τα κοινοβούλια των κρατών μελών είναι αυτά που έχουν στα χέρια τους την πραγματική δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεύτερον, θα πρέπει να κατανοήσουμε αλλήλους με καλύτερο τρόπο και την κοινή γνώμη μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό η συνεργασία μας πρέπει να γίνει πιο στενή. Και η ολοκλήρωση και ένταξη των κοινοβουλίων, των εθνικών, στους κοινοτικούς μηχανισμούς να γίνει με επιτυχέστερο τρόπο από ό,τι σήμερα. Ακούγονται πολλές ιδέες εδώ. Υπάρχουν πολλοί ε, εμπειρογνώμονες, πολύ περισσότερο από μένα σε τέτοια θέματα που αναφέρονται σε αυτό. Υπάρχουν νέες ιδέες για νέες κοινοβουλευτικές μορφές συνεργασίας, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί είναι ουσιαστικά μια στενότερη μορφή συνεργασία των κρατών μελών με την καθημερινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω κάποιων ιδεών που ακούστηκαν όπως η Επιτροπή Εθνικών Νομοθετών Έχει ήδη ακουστεί αυτό. Θα αποτελείται από μέλη των κρατών μελών και είναι το νέο σώμα το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν Συμβούλιο Επικρατείας, αν θέλετε, του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν περιπτώσει μπροστά μας έχουμε πάρα πολύ δύσκολες ε, εκλογικές διαδικασίες. Δεν είμαστε μόνοι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σε όλη την Ευρώπη νιώθουμε τον ευρωσκεπτικισμό να ανεβαίνει. Αυτοί που δεν εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά όργανα αυξάνονται. Αυτοί που θεωρούν ότι είναι δεδομένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, και νομίζω ότι οι εκλογές αυτές... Νομίζω ότι στις εκλογές αυτές θα πρέπει να αποσταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα από μας, από πλευράς μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες μας αγνοώντας τους πολίτες μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι πολίτες ψηφίζουν και για να ψηφίζουν πρέπει να εμπλακούν ακόμα περισσότερο στις διαδικασίες λήψης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το πετύχουμε. Thank you very much. Our next speaker... Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Βιτάλ Μοραέρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κάνω μια σύντομη παρέμβαση για το ρόλο των κοινοβουλίων, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων, σε θέματα εμπορίου, δυνάμει της παγκοσμιοποίησης. Το εμπόριο είναι ένας από τους πυλώνες της παγκοσμιοποίησης, όπως ξέρουμε και έχουμε πολύ περισσότερες εμπορικές συμφωνίες από ό,τι συμφωνίες σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι το πιο προηγμένο και εξεζητημένο σώμα διεθνούς διακυβέρνησης και παγκόσμιας διακυβέρνησης. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που ίσως ε, θα σας ε, καταπλήξει. Με μετά την ε, πρωινή παρέμβαση του κυρίου Τζόνσον δεν θα μπορούσε κανείς παρά να συμφωνήσει με αυτά που ακούσαμε ότι η ανάμειξη του, των κοινοβουλίων στην όλη διαδικασία και παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο. Γιατί δεν θα πρέπει απλώς ε, τα κοινοβούλια να κυρώνουν τις συμφωνίες ε, κατόπιν εορτής και αφού έχουν υπογραφεί από τις κυβερνήσεις, αλλά να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία από τα πιο πρώιμα στάδια. Γιατί από τη στιγμή που ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο θα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιήσουμε και τον τρόπο συμμετοχής ε, των εθνικών κοινοβουλίων στις διεθνείς σχέσεις γιατί οι διεθνείς σχέσεις δεν περιορίζονται πια μόνο στις εξωτερικές σχέσεις, στη διπλωματία, αλλά αφορούν τις μεταφορές, το κλίμα, το εμπόριο και πολλούς άλλους τομείς. Οπότε κάθε κεφάλαιο εθνικής διακυβέρνησης, κάθε τομέας εθνικής διακυβέρνησης έχει κάποια εξωτερική διάσταση. Οπότε τα εθνικά κοινοβούλια, αν θέλουν να ασκήσουν επιρροή και να επιδράσουν στις ε, πολιτικές σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εμπλακούν σε πρώιμο στάδιο και να συμμετέχουν στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, της διάφορες διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς. Θα σας ε, αφηγηθώ τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή την πρώιμη ε, συμμετοχή μας σε πρόωρο στάδιο της χάραξης της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ε, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε σκέφτεται είτε εξετάζει μια νέα διεθνή εμπορική συμφωνία, αποφασίζουμε και συντάσσουμε μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνήθως κάνουμε το ίδιο και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έρχεται στο Συμβούλιο και ζητά διαπραγματευτική εντολή. Έχουμε ήδη δηλαδή δύο εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, στην περίπτωση της ε, διατλαντικής εταιρικής σχέσης για εμπόριο και επενδύσεις, τη TIP, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεδριάσουμε δύο φορές. Μία πριν από κάθε, ε, την έναρξη κάθε γύρου διαπραγμάτευσης και μία μετά ώστε να γνωρίζουμε τι θα σκοπεύει να πει η Επιτροπή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να ενημερωθούμε και για την έκβαση του κάθε γύρω διαπραγματεύσεων. Επίσης, οργανώνουμε σεμινάρια, εργαστήρια, δημόσια κροάσεις, συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητήσεις με τους αρμόδιους επιτρόπους. Σε όλα τα στάδια λοιπόν των εμπορικών διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί πλήρη έλεγχο. Γι' αυτό και επιμένω και τονίζω αυτά που ακούσαμε το πρωί από τον Άντερ Τζόνσον. Αν θέλουμε πραγματικά να επιδράσουμε στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να ξεκινήσουμε ο καθένας στη χώρα του και στην Εθνική Βουλή να συμμετέχει στις διαδικασίες σε πρώιμο στάδιο. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και σε άλλους τομείς το εμπόριο πια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαράζεται και διαμορφώνεται από τα θεσμικά όργανα και όχι από τις ε, εθνικές κυβερνήσεις, ε, από εθνικά κοινοβούλια, αλλά αυτό μπορεί να ισχύσει για άλλους τομείς. Φυσικά, αν θέλουμε να λάβουμε μέρος στην παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει όλα τα κοινοβούλια να συμμετέχουμε σε διεθνή διακοινοβουλευτικά σώματα. Σε αυτά συμμετέχουν ε, εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές. Αλλά δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε με εθνικά ή δια, διακρατικά κοινοβούλια ε, ή κατηγορίες κοινοβουλίων που είναι διαφορετικές γιατί σε αυτές έχουμε άμεση εκλογή των μέλων. Εμείς ε, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική παγκοσμιοποίηση και σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε τρεις μορφές διεθνών διακοινοβουλευτικών σωμάτων. Ανάλογα με τους στόχους τους. Έχουμε διακοινοβουλευτικές ενώσεις που αφορούν κυρίως την διακοινοβουλευτική συνεργασία. Η IPU είναι η πιο παλιά διακοινοβουλευτική ένωση και πιο παγκοσμιοποιημένη τέτοια διακοινοβουλευτική ένωση, αλλά έχουμε και περιφερειακές διακοινοβουλευτικές ε, ενώσεις. Μερικές ε, είναι, στηρίζονται στη γλώσσα ή στηρίζονται στη θρησκεία ή μπορούν να έχουν οποιοδήποτε άλλο αίρισμα. Επίσης έχουμε διακοινοβουλευτικέ ενώσεις που θεσπίζονται μετά από διεθνείς συμφωνίες και παρακολουθούν την εφαρμογή και ελέγχουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμφωνιών. Στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πολλές διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν διακοινοβουλευτικό σώμα που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κοινοβουλίων των ε, συμβαλωμένων μερών της συμφωνίας. Στον τομέα του εμπορίου έχουμε το CARIFORM, που είναι διακοινοβουλευτική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των χωρών της Καραϊβικής, ε, που είναι από ανήκω χώρες ΑΚΕ και με τις οποίες έχουμε συνάψει εμπορική συμφωνία. Προβλέπεται επίση η σύσταση μια διακοινοβουλευτική επιτροπή που συμμετέχουν ευρωβουλευτέ και πρόσωποι βουλευτών των χωρών τη Καραϊβική και που παρακολουθούν την εφαρμογή αυτής της Διεθνούς Εμπορικής Συμφωνίας. Αυτά τα διακοινοβουλευτικά σώματα, επαναλαμβάνω, εξασφαλίζουν ένα follow-up αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Βέβαια, Αυτές είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε σε κάθε εμπορική συμφωνία συστηματικά την ίδρυση τέτοιου διακοινοβουλευτικού σώματος, όπως έχουμε με την Κάριφον. Για παράδειγμα, έχουμε μια ε, συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις δυτικοαφρικανικές χώρες και η συμφωνία αυτή δεν προβλέπει ε, σύσταση και ενό διακοινοβουλευτικού σώματος. Φαίνεται ότι άλλαξε πορεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θεωρεί ότι για την παρακολούθηση αυτών των διαπραγματεύσεων χρειάζεται συγκεκριμένο διακοινοβουλευτικό σώμα. Υπάρχουν όμω και κάποια διακοινοβουλευτικά σώματα που λειτουργούν ω συνελεύσει ή ω σώματα διεθνών οργανισμών. Για παράδειγμα, ανήκουν στο πλέγμα διακυβέρνησης ή στο σύστημα διακυβέρνησης διεθνών οργανισμών. Η πιο γνωστή περίπτωση και ε, μία από τις παλιότερες ε, περιπτώσεις και η συνέλευση με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη θέση παρατηρητή. Στον τομέα του εμπορίου τώρα, ένα παράδειγμα που θα ήθελα να λύσω κάπως πιο ενδελεχώς είναι η, η η συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, στην ε, Συμφωνία του Μαρακές το 1994 που δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν προβλεπόταν καμία διακοινοβουλευτική συνέλευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει συγκεκριμένους και πολύ αυστηρούς κανόνες και παρά τον σημαντικό ρόλο που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Εμπορίου ως σώμα που παράγει ε, κανόνες και νομοθεσία και έχει τέτοια λειτουργία, δεν υπάρχει παρόλα αυτά κοινοβουλευτική διάσταση στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η Διακοινοβουλευτική Ένωση, η IPU, αποφάσισε σε πολύ πρώιμο στάδιο να ξεκινήσει ένα είδος άτυπης κοινοβουλευτικής διάστασης ε, για το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και μας το ανέφερε αυτό το πρωί ο κύριος Τζόνσον. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία γιατί ιδρύθηκε έτσι όχι μόνο ένα μόνιμο όργανο με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και μάλιστα που συνέρχεται ετησίως, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία ε, διευθύνουσα επιτροπή που συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Έχουμε δύο συμπρόεδρου στην επιτροπή αυτή. Εγώ είμαι ο συμπρόεδρο εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο δεύτερο συμπρόεδρο εξασφαλίζεται από την Διακοινοβουλευτική Ένωση, την IPU. Εμεί προσδιορίζουμε το πρόγραμμα εργασιών τη ε, διευθύνουσα αυτή τη οι συνεδριάσεις γίνονται είτε στη Γενέβη είτε στις Βρυξέλλες. Η τελευταία έγινε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και επίσης ε, προσκαλέσαμε και τον Ρομπέρτο Σβίδλερ που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και συμμετείχε στη συνεδρίαση και τη Steering Committee της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΠΟΕ αλλά και στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή τη μας. Βέβαια, από την αρχή είχαμε την αντίθετη γνώμη όχι μόνο των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν κατά τη κοινοβουλευτική αυτή διάσταση του ΠΟΕ, γιατί δεν προβλεπόταν στι ιδρυτικέ συνθήκε του ΠΟΕ και επίση ε, θα επηρέαζε τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, των κυβερνήσεων ουσιαστικά, να αποφασίζουν από μόνε του για θέματα εμπορίου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα λοιπόν αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Χρειάστηκε μία δεκαετία για να υλοποιηθεί. Έτσι δημιουργήθηκε ένα, ένα σταθερό σώμα, προβλέψιμο με συμβουλευτικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα αναγνωριστήκαμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και γίναμε δεκτοί. Γιατί τώρα συνεδριάζουμε στα γραφεία του ΠΟΕ στη Γενέβη, κάτι που πριν από μια δεκαετία θα ήταν αδιανόητο, ασύλληπτο φέτος πια, τώρα πια γίνεται και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον Πασκάλ Λαμή το πρόεδρο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΠΟΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΕ. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή την ανυπαρξή επίσημη κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ με τη δημιουργία αυτή τη κοινοβουλευτική συνεργασία. Και αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για τη δημιουργία κοινοβουλευτικής διάστασης και σε άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Έθνη, το Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας ή το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Αυτά λοιπόν. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να έχουμε αντίκτυπο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον οίκο μας. Θα πρέπει να αλλάξουμε άρδιν τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας ε, και προσέγγισης ε, ε, της εκτελεστικής εξουσίας εκ μέρους των, Ευρωπαϊ... των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να συμμετέχουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, να τις κάνουμε εκτίμα μας και να, έχουμε συναντήσεις με την εκτελεστική μας ε, εξουσία και στη, κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και στην πορεία και κατά το τέλος των διαπραγματεύσεων. Αυτό το καταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον τομέα του εμπόριου και θα μπορούσε να, γίνει η δράση μας υπόδειγμα και για τα Εθνικά Κοινοβούλια για άλλους τομεί Έτσι θα εξασφαλίσουμε καλύτερη ανάμειξη των Εθνικών Κοινοβουλίων σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει η επιρροή μας και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί σε πολλές σημαντικές ε, διεθνείς οργανώσεις, όπως είπα, στα Ηνωμένα Έθνη, στη, στην Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας και το καθεξής, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτό δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει, θα πρέπει αντίθετα να ενδύνουμε τις προσπάθειές μας για να προσθέσουμε τέτοια κοινοβουλευτική διάσταση και σε παγκόσμιες οργανώσεις. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μπορώ να ξεκινήσω με λίγα λόγια για την κοινοβουλευτική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, πρώτου έρθω σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, της συνεδρίασής μας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με μία σειρά αξιών και αρχών. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η Επιτροπή Εξωτερικής ε, Δράσης, ως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ως το εκτελεστικό σώμα, φυσικά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου για τη δράση μας. Συγχρόνως όμως κατανοούμε ότι υπάρχει πολύ περιθώριο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα όπως είναι το θέμα που θα αποκαλούσα κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Τα κοινοβούλια, <clears throat> όπως είπα προηγουμένως, είναι υπέρμαχοι των αξιών, των αρχών, των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν περισσότερη ελευθερία κινήσεων από ότι οι εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν τους περιορισμούς που γνωρίζουμε όλοι. Επομένως μπορούν με πολύ χρήσιμο τρόπο να συμπληρώσουν τις δράσεις που αναλαμβάνονται είτε από τις εθνικές ε, διπλωματικές υπηρεσίες ή στη συγκεκριμένη περίπτωση από την ύπατη εκπρόσωπο και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Βλέποντας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπετε ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη γνώση σε σχέση με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς είδαμε ότι είναι τουλάχιστον 10 πρώην Πρωθυπουργοί και Υπουργοί Εξωτερικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι Ευρωβουλευτές και μπορούμε να αντλήσουμε από τη σοφία και τη γνώση τους. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος όμως, τι σημαίνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Για να παρουσιάσω ένα παράδειγμα το οποίο το γνωρίζετε όλοι, το θέμα της Ουκρανίας. Όλοι μας παρακολουθούμε τα γεγονότα, την προσπάθεια διαμεσολάβησης των Προέδρων Κόξ και Σαφνεύσκη, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είχαμε θαυμάσια σχέση μαζί τους. Αυτή η αποστολή βέβαια δεν είναι ενεργή τώρα, αλλά δεν έχει περατώσει πλήρω το έργο της για λόγους που είναι ανεξάρτητη τη θέλησή τους. Έχουμε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τους, δεν κάναμε καμιά προσπάθεια να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούν, αλλά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά μαζί τους και η αποστολή αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και υπό την έποψη του έργου της υπάτης εκπροσώπου και εμείς τους υποστηρίξαμε με κάθε τρόπο και με τη δική μας επιτόπια αντιπροσωπεία. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια και τα εθνικά επίση μπορούν να χρησιμοποιήσουν σημαντική θεσμική γνώση με χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση. Το έχουμε δει αυτό στο βόρειο τμήμα της Αφρικής, στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, όπου πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει εκ του μηδενό ένα σύστημα κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν να βοηθήσουν και να μεταλαμβαντεύσουν τι εμπειρίε του για το πώ μπορεί να οικοδομηθεί ένα σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου πάνω στην εκτελεστική εξουσία. Και το παράδειγμα <clears throat> το οποίο έρχεται στο μυαλό μου είναι φυσικά η Τινησία, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα επιτυχούς μετάβασης στη δημοκρατία. Τέλος, υπάρχει ο ρόλος τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινοβουλευτικοί στην παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών και αυτό είναι ένα κέριο εργαλείο εξωτερική πολιτικής από τη δική μας οπτική γωνία γιατί έχουμε μια εδρεωμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας όλες οι παρακολουθήσεις, όλες οι αποστολές ε, παρακολούθηση εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως ηγέτες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους προσδίδει αυτό και ανεξαρτησία αλλά και νομιμοποίηση στα μάτια των χωρών όπου γίνεται η παρακολούθηση των εκλογών. Δεν θα παραμείνω για πολύ στο θέμα των διεθνών κοινοβουλευτικών σωμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφερε πολύ καλά ο κύριος Μορέιρα. Ήθελα να τονίσω ότι και εμείς στην ε, γειτονιά μας έχουμε δύο κοινοβουλευτικά σώματα που ασχολούνται με τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις, η ΕΜΠΑ, η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και η λεγόμενη Euronest, η συνέλευση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία λοιπόν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και απαιτητική. Έχουμε τόσους πολλούς οι οποίοι εμπλέκονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις ε, εκτελεστικές υπηρεσίες, δηλαδή τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και εκεί η κύρια πρόκληση είναι να μπορέσει κανείς να έχει μια σωστή διαδικασία συντονισμού. Αναγνωρίζουμε βέβαια την ανεξαρτησία των κοινοβουλίων, την ανεξαρτησία του από οποιαδήποτε μορφή επιρροή που μπορεί να σκεφτεί από την εκτελεστική εξουσία. Συγχρόνως όμως είναι χρήσιμο να συνεννοούμεθα και να ανταλλάσσουμε απόψει για τα κύρια μηνύματα τα οποία δίδουμε. Όταν εγώ εργαζόμουν <clears throat> για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ, και αυτό έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων. Είτε πήγαινε στην Κίνα, είτε πήγαινε στην Αφρική. Τον άκουγαν όλοι οι συνομιλητέ του ω εκπρόσωπο της Ευρώπης. Γιατί για πάρα πολλούς δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον έξω κόσμο, για πολλούς είναι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ των απόψεων που εκφράσουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τη γνώση των ε, τοπικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αφρικανικές χώρες ή σε άλλες χώρες. Όταν μιλάμε λοιπόν για την κοινοβουλευτική διαδικασία και τη διάσταση την κοινοβουλευτική της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε και μια νέα εξέλιξη που είναι η διακοινοβουλευτική συνέλευση, κοινοβουλευτική συνέλευση για την ΚΕΠΑ, που είναι μια προσθήκη στην ΚΟΦΑΚ που είναι η συνέλευση των ε, Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και επίσης υπήρχε η αντίστοιχη Επιτροπή των Πρόεδρων των Επιτροπών Εθνικής Άμυνας των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων έχουν συγχωνευτεί τώρα αυτοί οι δύο φορείς και έχουν συγκροτήσει αυτή τη νέα Επιτροπή για την κοινοβουλευτική διάσταση της ΚΕΠΑ. Είναι ένα νέο εγχείρημα και η ύπατη εκπρόσωπος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ρόλο αυτού του φορέα και έχουν γίνει πολλές συναντήσεις από τότε που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αυτός ο νέος φορέας. Ξέρω ότι αυτή η κοινοβουλευτική συνέλευση για την ΚΕΠΑ δεν έχει επίσημα ελεγκτικά δικαιώματα και αρμοδιότητες, αλλά εμείς είμαστε σε επαφή μαζί τους, ακούμε τις απόψεις τους και έχουμε πάντα μια παρουσία στις ε, συνεδριάσεις τους σε υψηλό επίπεδο, είτε η ύπατη εκπρόσωπος, είτε υψηλή αξιωματούχοι. Είμαστε παρόντες λοιπόν στις συνεδριάσεις αυτού του σώματος και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια διαδραστικότητα, παραδείγματο χάρη με το να προσκαλούμε τους επικεφαλείς των αποστολών ΚΕΠΑ στους τομείς που συζητάει η συνέλευση αυτή. Αυτό είναι μια διαδικασία που μπορώ να παροτρύνω όλους να υιοθετήσουν. Αυτές είναι επιτυχείς λοιπόν διαδικασίες που ακολουθούν σε κάποιο βαθμό την κοινοβουλευτική ε, συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν, η οποία βέβαια πριν από δύο χρόνια καταργήθηκε πλήρως. Επομένω, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε και πολλά από τη συνεργασία με αυτή τη συνέλευση σε θέματα κέρια εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Τέλος, πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάν Βάουτερς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Οι διεθνείς οργανισμοί και οι μηχανισμοί διεθνούς διακυβέρνησης έμεσα αλλά και άμεσα επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι μια βασική διαπίστευση και θέτει το θέμα της παρουσίας και αντιπροσώπευσης και των δημοκρατικών εγγυήσεων. Ξέρουμε ότι οι διεθνείς οργανισμοί και τα διεθνή φόρα εν πολλής οργανώνονται από τις κυβερνήσεις. Αυτές οι οργανώσεις και τα φόρα αυτά στην ουσία πολλές φορές λειτουργούν σαν λέσχες της εκτελεστικής εξουσίας. Πρόκειται για μια αρπαγή, αν θέλετε, της εξουσίας στα πλαίσια της πολυμερούς διπλωματίας. Αυτή, αυτός είναι ένας όρος ο οποίος είναι, θα έλεγα, στο εσωτερικό μας, στο άρθρο 21 της συνθήκης. Αλλά αυτή η πολυμέρεια της διεθνούς σκηνής και των διεθνών σχέσεων στην ουσία δεν είναι παρά μία λέσχη πολύ κλειστή όπου ισχυρές χώρες συναντώνται, πολλές φορές ε, οι χώρες αυτές ε, έχουν δικαίωμα είτε νομικό είτε έμεσα κυρίαρχο ε, βέτο στις λέσχες αυτές. Η εξουσία αυτών των οργανώσεων είναι, θα έλεγε κανείς, σχετικά περιορισμένη. Κάποιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν φυσικά κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, Είδαμε παραδείγματα το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, ο ΑΣΕ λοιπά. Οι αρμοδιότητες αυτών των κοινοβουλευτικών σωμάτων είναι άνισες μεταξύ τους. Και πολλές φορές στο παράρτημα τουλάχιστον που έχουμε μπροστά μας μπορείτε να συγκρίνετε το τι κάνουν αυτές οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Έχουμε και την IPU, είδαμε και τον εκλεκτό γενικό γραμματέα της σήμερα, που υπερασπίζεται φυσικά τα κοινοβουλευτικά δίκτυα, την διεθνή διάσταση του κοινοβουλευτισμού. Πέραν αυτού όμως η IPU δεν είναι κάτι το οποίο συνδέεται επίσημα με ένα θεσμικό ε, σύνολο οργανωτικό. Δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει για να γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι δεν υπάρχουν πραγματικά διακυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες να έχουν ενσωματωμένη κοινοβουλευτική διάσταση. Τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται με την IPU, αλλά δεν έχουν ουσιαστικά κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτό το είπε και ο Γιώ νωρίτερα. Υπάρχει μια κίνηση για να υπάρξει μια διακοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά η υποδοχή της πρότασης αυτής είναι χλιαρή από τους περισσότερους υπουργούς εξωτερικών και διπλωμάτες. Υπάρχουν και άλλες λιγότερο θεσμικές μορφές συνεργασίας όπως οι G8, οι G20 που έχουν κάποιες διαστάσεις κοινοβουλευτικές με τη μορφή της συνάντησης των προέδρων των κοινοβουλίων τους, αλλά δεν επηρεάζουν και ιδιαίτερα τις διαδικασίες λήψης απόφασης που λαμβάνονται πάντα από, τις, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και αγνοούν πολύ στην κοινοβουλευτική διάσταση. Λόγω αυτής της υποανάπτυκτης κοινοβουλευτικής διαδικασίας αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί προβλήματα, προβλήματα εμπιστοσύνης, διαφάνειας, ευθύνης, λογοδοσίας και σύνδεσης με τις προσδοκίες των πολιτών. Τι μπορούμε να μάθουμε στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης και πράγματι έχουν υπάρξει και με τη συνθήκη της Λισαβόνας κάποιες προσθήκες της κοινοβουλευτικής διάστασης στις κοινοτικές αρμοδιότητες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της κοινή εμπορικής πολιτικής. Είδαμε μια θεσμοποίηση και ενίσχυση της, ε, σε μεγάλη διάρκεια πλέον εμπλοκής των κοινοβουλίων των κρατών μελών και είδαμε επίσης και αυξημένα παραδείγματα της IPC, της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει από την Κοζάκ, πολύ γνωστή, από την διάσκευση IPC για την ΚΕΠΑ όπως επίσης την διάσκεψη IPC για οικονομική διακυβέρνηση που προβλέπεται από, τη συνθήκη, από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Συνεργασίας της Ευρωζώνης κτλ. Υπάρχουν και αρκετές συναντήσεις ad hoc IPC σε θέματα που επιλέγουν τα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει και ο μηχανισμός προστασίας της αρχής της επικουρικότητας τι, εμπειρία έχουμε από όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι κάτι χρήσιμο, μπορούμε να το συστήσουμε και σε άλλα διεθνή επίπεδα συνεργασίας. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτοί οι μηχανισμοί IPC δεν έχουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων. Εμπλέκονται βέβαια και αναπτύσσονται με ευέλικτο τρόπο και εμπλέκονται επίσης και σε κάποιες ουσιαστικές δημοκρατικές λειτουργίες. Δεν θα εξαντλήσω τον κατάλογο αυτό τώρα, αλλά ασχολούνται με θέμα ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, διεκτύωσης, των think tank. Ξέρετε ότι είχαμε ε, μια διάσκεψη στο παρελθόν ε, μια συνάντηση κοινοβουλευτική και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο ΚΟΖΑΚ και νομίζω ότι τα think tanks είναι αρκετά χρήσιμα και αυτά γιατί οι βουλευτές μέσα από αυτά μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους περίπλοκα στοιχεία, δεδομένα και να αποκτούν μερικές φορές ευρύτερες προοπτικές από ότι οι υπεύθυνοι κάθε φορά των δημοσίων υπηρεσιών με τις οποίες συνεργάζονται. Προσπαθούμε να είμαστε πράγματι, ε, αν θέλετε, εμπλεκόμενοι στην διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή η οποία κυριαρχείται από τις κυβερνήσεις ακόμα περισσότερο στον τομέα της ΚΕΠΑ και τα λοιπά και φυσικά της άμυνας. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα που άπτονται τη πανεπιστημιακής έρευνα, σαν παράδειγμα. Σε επίπεδο πολιτικό-φιλοσοφικό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι τα κοινοβούλια και οι κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί παρέχουν το πλαίσιο, το φόρουμ, στο εσωτερικό του οποίου μπορεί να εξελιχθούν πολιτικές συζητήσεις που να γίνουν ορατές στους πολίτες να δουν οι πολίτες ότι υπάρχει χώρος, χώρος συζήτησης, χώρος αμφισβήτησης, χώρος εναλλακτικών προτάσεων πέρα από τις καθιερωμένες πολιτικές εκφράσεις. Είναι βασική λειτουργία των κοινοβουλευτικών μηχανισμών. Τι μπορούμε να μάθουμε τώρα λοιπόν από τις εμπειρίες αυτές για τους διεθνείς τουλάχιστον οργανισμούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε <clears throat> είναι καταρχάς το εξής. Θα βρείτε άλλωστε στο τέλος της αίθουσας ε, κάποια αντίγραφα ενός σημειώματος που έγινε διαθέσιμο από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, προχωρημένη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά εξηγούν θα έλεγα ε, με σωστό τρόπο ε, το πώς λειτουργεί η διαδικασία IPC. Και τι βλέπει κανείς αυτά τα σημειώματα. Βλέπουμε ότι με την σόρευση αυτών των σωμάτων IPC, κοινοβουλευτική συνεργασίας, στην ουσία πέφτουν θύματα της ίδια τους της επιτυχίας. Έχουν πάρα πολύ παραφορτωμένες ημερήσιες διατάξεις Οικονομικά είναι δύσκολο τα μέλη των κοινοβουλίων να ταξιδεύουν δεξιά και αριστερά και ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο ε, δεν πετυχαίνει τους στόχους του, διότι λόγω ακριβώς του μεγάλου αριθμού των φόρα αυτών υπάρχει μια διάχυση ενέργειας και υπάρχει μια κόποση, μια αίσθηση κόπωσης αυτών των μορφών κοινοβουλευτική συνεργασίας. Ε, έγινε μια έκθεση πρόσφατα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου που λέει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθούν και να οργανωθούν σοβαρά έτσι ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και να δοθεί μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα κλείσω τώρα πρόεδρε, θα σας πω ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση μπορεί να βελτιωθεί και να επωφεληθεί από τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μια πολυδιάσπαση του κοινοβουλευτικού στοιχείου. Αν γίνει μια υπερβολική εξειδίκευση του κοινοβουλευτικού στοιχείου, τότε θα γίνουμε αυτό που ονομάζεται talking shop, δηλαδή απλά έτσι σημεία κουτσομπολιού ας πούμε. Και δεν θα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των κοινοβουλευτικών. Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί ο αριθμός των συναντήσεων IPC, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνουμε τα, κράτη των κοινοβου... τα μέλη των κοινοβουλίων να πηγαίνουν κάπου λόγω ε, της σύμπτωσης πολλών συναντήσεων και του οικονομικού βάρους. Κάνουμε πολλές μελέτες στα πλαίσια της μελέτης μας και είδαμε ότι οι μηχανισμοί IPC είναι αρκετά ικανοί να μην συζητούν αφηρημένες τομείς, ε, γενικά όπως ας πούμε η αλλαγή του κλίματος, αλλά να ασχολούνται με πολύ συγκεκριμένα επικεντρωμένα θέματα. Αυτό είναι ένα κίνητρο για τους βουλευτές να εμπλέκονται και να ενδιαφέρονται. Με άλλα λόγια, το βασικό επιχείρημά μου ποιο είναι. Είναι μεν ενδιαφέρον να θεωρήσει κανείς το παράδειγμα των IPC σαν ένα καλό παράδειγμα, να δούμε μουτά της μουτάντης εάν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο το ευρωπαϊκό, από τη λειτουργία τους, αλλά να παραμείνει περιορισμένος ο αριθμός αυτών των φόρα, και να συναντώνται οι κοινοβουλευτικοί που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα και να παίζουν τον δημοκρατικό τους ρόλο ο οποίος τους έχει αποδοθεί και αποτελούν πράγματι ένα αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Έχω τρεις ομιλητές τώρα που θα λάβουν το λόγο. Ο πρώτος μας ομιλητής λοιπόν. Ο κ. Μάρκ Έλσιολ από το Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο ως πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου. Εμείς είμαστε ένα μικρό κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι ε, κατά την άποψή μου όλοι μας δεν πρέπει να ξεχνάμε είτε είμαστε από μικρά είτε από μεγάλα κοινοβουλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση στα κοινοβουλιά μας. Και πέρα από αυτήν την ευρωπαϊκή διάσταση, αυτό που συζητάμε σήμερα, αυτό που πρέπει να ε, μην ξεχνάμε είναι ότι οι Βρυξέλλες ε, δεν είναι μακριά. Αυτή είναι μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Και πρέπει να σα πω ότι στην αρχή λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συνάδελφοι ε, που έχουν ε, ευρωπαϊκές προτάσεις για την επικουρικότητα και μετά όταν ψηφίζουμε λένε ξαφνικά «Μα δεν έχω ακούσει τίποτα». Άρα δηλαδή ας μην το ξεχνάνε αυτό οι συνάδελφοί μας. Το δεύτερο θέλω να πω σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Μπάουτσα, αν τον κατάλαβα καλά, είναι, μας είπε ότι ορισμένα ε, διακοινοβουλευτικά ε, φόρα παίζουν το ρόλο της ε, δεξαμενής ταλέντων και σοφών. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την συνέλευση που έχει μια πολύ καλά λειτουργούσα γραμματεία εγώ ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ως βουλευτή να έρθω σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό κόσμο, με την κοινωνία των πολιτών, με ΜΚΟ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό. Δηλαδή, από την κοινοβουλευτική του δουλειά ε, επιλέγει κανείς αυτά που αφορούν τις ΜΚΟ ε, και άλλους παρεμφερείς οργανισμούς. Και κάτι άλλο. Ε, όταν αποκτήσει κανείς ε, περισσότερη εμπειρία, ε, του ζητούν να εκπροσωπήσει ένα κοινοβουλίο και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Γιατί δεν πρέπει να σαντά κανείς πάντα τους ίδιους ανθρώπους, να υπάρχει κατανομή εργασίας, να αφήσουμε και τους συναντέλφους μας να αποκτήσουν εμπειρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια πρέπει να το λέω και στον εαυτό μου. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αποκτήσουν αυτή την ε, ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση στην ε, καθημερινή του ζωή ως βουλευτές. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ενισχυμένη συνεργασία και επαφές με τις άλλες ειδικευμένε επιτροπές. Και φυσικά υπάρχει η συνάντηση της ΚΟΖΑΚ, υπάρχει η Επιτροπή για την ΚΕΠΑ, όλα αυτά είναι επιτροπές οι οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα κοινοβουλευτικά θέματα, όπως και η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πάντα θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε την ε, αντιπροσώπευση και των ε, αρμοδίων επιτροπών. Η πολιτική η ευρωπαϊκή δεν είναι μονάχα εξωτερική πολιτική, είναι μια πολιτική που ενδιαφέρει όλους τους τομείς. Φυσικά είναι χρήσιμο να λάβει κανείς υπόψη την ανάγκη να υπάρχουν από τους εκπροσώπους οι κατάλληλες γλωσσικές ικανότητες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πάντα ο ρόλος της συναπόφασης σε όλες αυτές τις ε, ε, διοργανώσεις. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην Άννα Γκάμισ. Α, εδώ είσαστε, είσαστε παρούσα. Ε, ευχαριστώ. Ε, καταλαβαίνω αυτά που είπε ο καθηγητής Βόουτερς ότι δηλαδή δημιουργείται μια κόποση των κοινοβουλευτικών διασκέψεων. Και εγώ φοβάμαι ότι είχαμε μεγάλο αριθμό κοινοβουλευτικών φόρουμ. Γιατί με τέτοιο κοινοβουλευτικό τουρισμό δεν θα κερδίσουμε και πολλά. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνεχώς επαφές με την κοινωνία των πολιτών, με think tanks, από αυτή την άποψη λοιπόν θα έλεγα ότι στη διάσκεψη αυτή μιλάμε για τα Εθνικά Κοινοβούλια και την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και δεν μπορούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο να ξεχνούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη και την έδρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι αναπόφευκτο ένα τέτοιο θέμα. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας με μία έδρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αυτονόητο σε μία παγκόσμια διακυβέρνηση. Και αν δεν το θέσουμε εμείς αυτό το ζήτημα, ποιος το θέσει. Είναι δικό μας καθήκον και έργο. Και σίγουρα χρειαζόμαστε καλύτερη διάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και για την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας. Και εκεί σίγουρα υπάρχει πρόοδος με τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη και τις τακτικές μας επαφές. Για παράδειγμα, εμείς επισημάναμε στους εθνικού βουλευτές που δεν το γνώριζαν το αίτημα μας να αναθεωρηθούν οι μηχανισμοί για την χρηματοδότηση των αποστολών κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Γιατί ο ισχύων μηχανισμός όχι μόνο είναι άδικος, αλλά είναι και αναποτελεσματικός. Γιατί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιες δυνάμεις για να προστατεύσουμε τις αποστολές μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και απασχίζουμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί ο μηχανισμός χρηματοδότησης των αποστολών της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μας δεν χειροπόδαρα αντί να διευκολύνει την ανάληψη δράσεων. Θέλουμε λοιπόν καλύτερο συντονισμό με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική, ε, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Εξωτερικών Ασφάλεια και Άμυνας. Και επίσης θέλουμε καλύτερο συντονισμό και με την ΕΕΔ, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά και καλύτερη συνεργασία και επαφή με το Συμβούλιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που έχουμε με συνεπή συγκροτημένο τρόπο για την ανάπτυξη του εμπόριο, την ενέργεια, ανθρωπιστικά θέματα, ανθρωπιστική πολιτική, στην πολιτική γειτονία και ούτω καθεξής. Λείπουν αυτά τα στοιχεία. Αναφέρθηκαν κάποια επιτυχή σενάρια, κάποιες επιτυχείς πρωτοβουλίες, τα θέματα της Τινησίας και της Ουκρανίας. Εκεί ήταν επιτυχημένη η παρέμβασή μας. Αλλά είχαμε και αρνητικές περιπτώσεις, πολύ απογοητευτικές, με ολέθρια αποτελέσματα. Συρία, Λιβύη για παράδειγμα. Δυστυχώς η κατάσταση στη Συρία είναι χαοτική. Είναι παταγώδης αποτυχία εξαιτίας έλλειψης συντονισμού. Όχι μόνο σε επίπεδο ΑΕΔ, αλλά και σε επίπεδο χωρών μελών. Δυστυχώς δεν υπήρξε συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και παρά την θετική αντίδραση της Λιβύης και εκεί είχαμε καταστροφή. Και σίγουρα η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω πριν αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια βελτίωση. Και εμείς φταίμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρλος Κωνστανέβες από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να είμαι σε αυτήν την ε, συνεδρίαση. Αγαπητέ Όθμαρ, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους και θα ήθελα να τονίσω πόσο χαίρομαι που είμαι πάλι σε αυτή την αίθουσα που παλιά ήταν η αίθουσα των συνεδριάσεων της πολιτικής μου ομάδας και με νοσταλγία επανέρχομαι εδώ για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Εγώ με την άποψη ότι αυτή είναι μια χρήσιμη συνεδρίαση, μια εύστοχη συνεδρίαση και πρέπει να θεωρηθεί ότι όλες αυτές οι ανησυχίες που τρέφουμε όλοι μας, ο πολλαπλασιασμός, η πολυπληθώρα των συνελεύσεων και των συναντήσεων, οι διεθνείς αυτές σχέσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ότι αυτό καθώς και η ανάγκη να υπάρχει καλύτερη διαδικασία συντονισμού και συνάρθρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Είναι λοιπόν και μια ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε αμοιβαίο εμπλουτισμό γνώσεων σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Πορτογαλία εμεί έχουμε ιδιαίτερου λόγου να θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ήμασταν πάντα μια χώρα γέφυρα κατά κάποιο τρόπο και έχουμε κάποιες εμπειρίες που μπορούμε να μεταλαμβαδεύσουμε και σε άλλους που μπορεί να είναι χρήσιμες. Εμείς λοιπόν ως Εθνικά Κοινοβούλια, ως Εθνική Κοινοβουλευτική, ε, εγώ συγκεκριμένα ως ένα άτομο που πέρασε από το Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κυβέρνηση της χώρας μου, Νομίζω ότι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους ενός κοινοβουλίου είναι να μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί τη δράση μιας κυβέρνησης στους διεθνείς φορείς. Να παρακολουθεί λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει όχι μονάχα το... η κυβέρνηση μιας χώρας, αλλά το ίδιο ισχύει και για το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς λειτουργούν διάφοροι σχηματισμοί του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση, να την χάνουν μεγαλύτερες παρακολούθησης και μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού ελέγχου από τα εθνικά τους κοινοβούλια και ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά όπου εμπλέκονται ευρωπαϊκά θέματα και εξωτερικές σχέσεις. Όταν πρόκειται τώρα για την ε, μορφή με την οποία θα γίνει αυτή η σύνδεση, Όλοι μας σκεφτόμαστε ένα ιδανικό σχήμα. Θα θέλαμε να ήταν πράγματι πολύ στενή η σχέση των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει μια βαθιά συνεννόηση και διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών. Εμείς έχουμε ε, πολλές συνεδριάσεις οι οποίες έχουν διοργανωθεί με αυτό το στόχο. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε πετύχει ακόμα το ιδανικό σχήμα για αυτή τη συνεργασία. Για τα θέματα λοιπόν που συζητούμε σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει μια απαρχή, μια εκκίνηση η οποία φαίνεται σε ορισμένου ότι δεν είναι ίσως αρκετά φιλόδοξη, αλλά θα μπορούσε να είναι επωφελής αν όλα τα εθνικά κοινοβούλια έπαιρναν από το, Εθνικό Κοινο... από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγγνώμη, τις ε, εντολές που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διεθνείς σχέσεις, Τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορούμε να γνωρίσουμε εκ των προτέρων ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε να συζητούμε κατά πόσον συμφωνούμε ή όχι με μια τέτοια προσέγγιση. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόταση για ένα πρώτο βήμα που δεν είναι παρά μόνο <clears throat> ένα απλό βήμα χωρίς τρόμενες φιλοδοξίες αλλά μπορεί να είναι μια πολύ καλή αρχή. Και θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την άποψή μου σε σχέση με το επόμενο θέμα που θα συζητηθεί, που είναι μια κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Όπω είπε και η συνάδελφό μου, η Άννα έχουμε εδώ μια μεγάλη πρόκληση για το πώς θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Είτε εγκαταλείποντας τι εθνικέ εκπροσωπήσει ή δουλεύοντα παράλληλα με αυτέ τι εθνικέ αντιπροσωπείε. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε και για μια άμεση εκλογή των βουλευτών που θα συμμετέχουν στην ε, συνέλευση αυτή των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ένα τέτοιο βήμα, να έχουμε μια συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που να απαρτίζεται από εθνικούς κοινοβουλευτικούς, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε καν αρχίσει να επιτυγχάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά καταρχήν σας ε, καλωσορίζουμε που επανήλθατε. Η κυρία Γκαμπριέλε Κρετή είναι η τελευταία που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι επιστημολόγος και όμως είμαι και δημοκράτης και γι' αυτό ε, ξέρω πολύ καλά ε, ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε προβλήματα που δεν έχουν διατυπωθεί καλά και κανένας ε, πολίτης δεν θα βρει μία απάντηση απλά και μόνο υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί οποτεδήποτε πρόκειται για την δημιουργία δημοκρατικού πλαισίου όπου μεταβιβάζουμε την ευθύνη σε οργανισμούς που δεν είναι δημοκρατικοί και όταν προσπαθούμε να ασκήσουμε έλεγχο και να παραμείνουμε ενημερωμένοι. Εάν λοιπόν θέλουμε να καλέσουμε κάποιον να λογοδοτήσει, είναι σαν να προσδίδουμε νομιμοποίηση εκ των υστέρων. Όμως η νομιμοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει μόνο για την, με την ανάληψη ευθυνών για αυτά τα οποία πράττουμε. Η νομιμοποίηση έχει σχέση και με το στόχο. Και νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε ευθύνες για κάποιες ε, πολιτικές ε, που είναι λάθος. Μερικές φορές και οι στόχοι είναι λάθος. Ε, χάρη πρέπει να δούμε λιγάκι τις πολιτικές λιτότητας στην Ευρώπη αν οι πολιτικές αυτές ε, δεν γίνονται αποδεκτές, αυτό όχι διότι δεν πέρασαν από το Κοινοβούλιο, αλλά ε, διότι ορισμένα μέτρα ήταν ευθύς εξ αρχής ε, λανθασμένα. Γιατί λοιπόν να πρέπει να νομοποιήσουμε κάποια μέτρα που δεν ήταν καλά ευθύς εξ αρχής. Ο δικός μας ο στόχος είναι να επιλέξουμε αυτό που είναι καλύτερο στην κοινωνία που ζούμε. Και αν αυτό μπορεί να εγκριθεί, τότε θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει το ρόλο μας και ο ρόλος μας, ε, το άσχημο στο ρόλο μας ήταν ότι ήμασταν αποκλεισμένοι όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά πολλές φορές και σε εθνικό επίπεδο. Και ορισμένοι είπαν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει διαφάνεια, ε, να προσφέρονται πληροφορίες, να υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Άρα δηλαδή ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι βουλευτές κατά κάποιον τρόπο ε, να λειτουργούν ως μάνατζερ και εάν είσαστε ευχαριστημένοι με αυτό ε, τότε θα πρέπει να ερμηνεύσουμε σωστά το ρόλο μας. Και οι βουλευτές είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι απλά δεν θα έχουν πια εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Συζητήσαμε διαμακρών τι ρόλο ε, πρέπει να διαδραματίσουμε σχετικά με τις ε, δαπάνες του προϋπολογισμού. Εάν το ευρωπαϊκό εξάμεινο προβλέπει ότι πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένα μέτρα και ορισμένες ε, κυβερνήσεις ε, δέχονται αυτά τα μέτρα ε, χωρίς καμία εξαίρεση, τότε αυτός που έχει να χάσει είναι το Κοινοβούλιο. Εκείνο χάνει, διότι κατ' ουσίαν είναι μία δύναμη μέσα στην αδυναμία. Και δεν θέλω πια να φιλοσοφήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως θέλει κάποιος από τους ομιλητές να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε Μορέιρα. Έχω μερικές επιπλέον παρατηρήσεις για να εμπλουτίσω και την αρχική μου ομιλία. Σήμερα δεν είναι θέμα μας η ενδοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική συνεργασία. Θέμα της σημερινής διάσκεψης είναι η συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή εκτό των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και πολλές παρατηρήσεις ε, που ακούσαμε και το πρωί και το απόγευμα ήταν λίγο εκτός θέματος. Ας ε, εμείνουμε λοιπόν στο κυρίως θέμα της σημερινής μας συνάντησης. Σε ορισμένους τομείς για τους οποίους ισχύει κοινοτική αρμοδιότητα, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για παράδειγμα, δεν είμαστε μέλη των βασικών διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας και άμυνας, δηλαδή ΝΑΤΟ, ε, Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΙΕ ή Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ. Δεν είμαστε μέλη στις διεθνείς αυτές, στις διεθνείς αυτές οργανώσεις και οργανισμούς. Τα κράτη-μέλη είναι μέλη αυτών των διεθνών οργανώσεων. Υπάρχουν όμως ε, κανόνες και διατάξεις της συνθήκη της Λισαβόνας που ρυθμίζουν αυτό το θέμα της ε, συμμετοχής σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων που αναφέρουν ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για θέματα εξωτερικής πολιτικής όταν αυτές ε, υπάρχουν. Οπότε, τα κράτη-μέλη που είναι μέλη σε διεθνείς οργανώσεις ε, δεσμεύονται στις θέσεις τους εκεί από τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχουμε όμως διακοινοβουλευτικές οργανώσεις, τότε είναι τα εθνικά κοινοβούλια που θα πρέπει να δώσουν το παρόν εκεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος σε τέτοιες διακοινοβουλευτικές οργανώσεις. Και εκεί τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας διάστασης. Έχουμε όμω άλλου οργανισμού ή άλλε οργανώσεις στους οποίους ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ηδη η επίση μέλο, παράλληλα με τα κράτη-μέλη, όπως στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν ξέρω γιατί τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφόσον ε, η εμπορική πολιτική είναι πια αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτόνομο μέλος του ΠΟΕ. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούν και τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, είναι μέλη στη ΦΑΟ, στο πρωτόκολλο του Κιώτο και σε άλλες οργανώσεις, όπως στον ενεργειακό χάρτη. Έχω ολόκληρο κατάλογο εδώ με διεθνείς οργανώσεις. Δεν χρειάζεται να σας τον διαβάσω. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν να είναι μέλη διακοινοβουλευτικών σωμάτων που προβλέπονται στις συνθήκες αυτών των οργανώσεων. Έχουμε μερικέ περιπτώσει όμω που μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλο τέτοιων οργανώσεων, όπω στην Παγκόσμια Τελωνιακή Ένωση. Εκεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλο τη Παγκόσμια Τελωνιακή Ένωση. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αυτό όμως δεν ισχύει ακόμη. Οπότε, σε θεσμοθετημένη συμμετοχή είναι συγκεκριμένε οι περιπτώσεις που μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει. Τώρα, όταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι μέλη των συνθηκών ή των οργανώσεων, τότε και οι δύο φορείς ε, δικαιούνται να αναπτύξουν την κοινοβουλευτική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προβλέψουμε μηχανισμούς για να συντονίσουμε τη συμμετοχή μας σε τέτοιες διεθνείς οργανώσεις και φόρα. Όταν όμως μόνο τα κράτη-μέλη είναι μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να ενισχύσουν αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση, έχοντας κάνει ένα συντονισμό μεταξύ τους. Γιατί σε τέτοια περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει σε τέτοιε οργανώσει, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλο μια διεθνή οργάνωση μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διάσταση τέτοια οργάνωση. Οπότε έχουμε πολύ έργο μπροστά μα και θα πρέπει όχι μόνο να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα συμμετέχουμε και πώ θα ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση διεθνών οργανισμών, αλλά και θα πρέπει να δούμε πώ θα συντονιστούμε μεταξύ μα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια, όταν και εμεί και εσεί δικαιούμαστε να συμμετέχουμε στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Στην περίπτωση του ΠΟΕ, ακριβώς επειδή τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να είναι μέλη του ΠΟΕ, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Γιατί και τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Ένωσης και συμμετέχουν και στην Διεθνούς Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΠΟΕ. Οπότε και ο άλλος συμπρόεδρος της, ε, του Steering Committee είναι Ευρωπαίος. Οπότε αυτή τη στιγμή και οι δύο συμπρόεδροι της Διευθύνωση Επιτροπής της κοινοβουλευτική Συνέλευσης του ΠΟΕ είναι Ευρωπαίοι. Είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Είναι Ευρωπαίοι βουλευτές. Εγώ ως ευρωβουλευτή και ο Σουηδό συνάδελφος είναι Σουηδό βουλευτής. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε την ύπαρξη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για να συνδυάσουμε και να συντονίσουμε τη συμμετοχή μας και να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Γιατί αν υπάρχει υπερβολικός κατακαιρματισμός θα έχουμε πολλαπλασιασμό των κοινοβουλευτικών διασκέψεων και περιττή επανάληψη και επικάλυψη. Και διατρέχει ο κίνδυνος να γίνουμε πλανώδη βουλευτές, πλανώδη κοινοβουλευτικοί. Κάτι που θα αμαυρώσει την εικόνα των κοινοβουλίων στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Ας μην ξεχνάμε και αυτό το κίνδυνο λοιπόν. Η κυρία Μπακογιάννη. Ε, φοβάμαι ότι εγώ δεν το είχα καταλάβει σωστά το θέμα. Εγώ είχα καταλάβει ότι θα μιλάγαμε για το πώς τα εθνικά κοινοβούλια θα διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο την διαδικασία την ευρωπαϊκή και τη διαδικασία της παγκοσμιοποίηση. Εγώ έτσι είχα καταλάβει. Αλλά τελικά φοβάμαι ότι όλη η συζήτηση έγινε πάρα πολύ τεχνική και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό που κατά τη δική μου άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό τώρα είναι το πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψουμε στους πολίτες. Και το πολιτικό αυτό μήνυμα ε, δεν έχει σχέση με το ταξιδεύουμε πολύ, αν έχουμε ε, πολλούς οργανισμούς, αν συναντιόμαστε στο Τόκιο ή στις Βρυξέλλες, αν ε, συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού σε ποια κοινοβουλευτική συνέλευση. Σήμερα δεν τίθεται αυτό το ερώτημα και νομίζω ότι τελικά ε, πολλοί στην Ελλάδα τουλάχιστον πολλοί κάθονται πολίτες και συζητάνε ε, μάλλον δεν συζητάνε για το αν ένας βουλευτής συμμετέχει ή όχι σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό που θέλει ο πολίτης είναι το κατά πόσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται και είναι σημαντικές για το μέλλον, δεν θα τον επηρεάσουν άμεσα ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να διαδραματίσουν πιο σημαντικό ρόλο. Είμαι απόλυτα πεπισμένη για τον ε, ε, αποτελεσματικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ, εντάξει, μέχρι τώρα ήμουν ή μέλος κυβέρνησης ή βουλευτής και έκανα τελείως διαφορετική δουλειά από αυτή που κάνετε εσείς. Όμως, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός ο οποίος είναι κοντά στους πολίτες. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα μεταφέρουμε στους πολίτες, να τους κάνουμε να κατανοήσουν και φοβάμαι ότι τελικά μιλάμε διαφορετική γλώσσα στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κατά κάποιον τρόπο ίσως αυτό να είναι φυσιολογικό. Όμως ε, μία επαφή, μία πιο άμεση επαφή είναι πραγματικά απαραίτητη. Και ε, τώρα μιλάω εκ μέρους της ε, ε, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τα κοινοβούλια, αλλά τα κοινοβούλια είναι υπόλογα απέναντι στους πολίτες. Άρα δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε Κοιτάξτε, δεν έχω να σας παρουσιάσω τώρα κάποια συγκεκριμένη πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερα φόρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οι αποφάσεις να λαμβάνονται διαφορετικά. Η εθνική, ε, τα εθνικά κοινοβούλια και η εθνική πολιτική να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι μέχρι τώρα. Οι βουλευτές να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων. Και αυτήν την ε, απάντηση να τη βρούμε το στομότερο δυνατόν, το αργότερο ε, μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές και οι προτάσεις αυτές να παρουσιαστούν από τα κόμματά μας. Διότι υπάρχει το κενό, αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός υπάρχει, η παγκοσμιοποίηση, οι άνθρωποι βιώνουν μόνο την αρνητική πλευρά της παγκοσμιοποίησης, άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο συγκεκριμένες ε, ε, ιδέες. Και ξέρετε, ε, ελπίζω τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές να είμαστε περισσότερο έτοιμοι να καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις που είναι απαραίτητες. Και κλείνω λέγοντας ότι τελικά φοβάμαι θα πρέπει να βρούμε κοινή γλώσσα. Λιγότερο τεχνική. Συγγνώμη τώρα αν ε, χρησιμοποιήσω λάθος λέξη, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λιγότερο γραφειοκρατική, λιγότερο τεχνοκρατική και περισσότερο πολιτική, αν θέλουμε πραγματικά να περάσουμε ένα μήνυμα στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει ένας υπερβολικός αριθμός σωμάτων και είναι δύσκολο να τα εξυπηρετήσει κανείς μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να τα εγκαταλείψει από κάποια στιγμή. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ώσπου να ενσωματωθεί το κοινοβουλευτικό σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επανέλθω σε αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Μορέιρα στα ήδη υπάρχοντα κοινοβουλευτικά σώματα, οι βουλευτές είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσουν να λειτουργούν σαν ένα ευρωπαϊκό σύνολο, σαν ένα ευρωπαϊκός πυρήνας. Το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος ή όχι του συγκεκριμένου οργανισμού είναι κάτι που μας διευκολύνει εφόσον είναι βέβαια να μεταφέρουμε το κοινό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε σαν ενδιάμεση. Σαν παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα θέματα μετα... και στο... στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΑΣΕ για θέματα εκλογικών διαδικασιών σε άλλες χώρες. Και εδώ τα κοινοβούλια τα εθνικά που είναι και στις δύο πλευρές μπορούν με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν διαιτητικά αν θέλετε διαμεσολαβώντας. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά. Στον τομέα που εργάζομαι εγώ υπάρχουν κάποιες διαφορές συχνά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Πολλά προτείνονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε στα δικά μας μέλη. Υπάρχουν απορίες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα θέματα κάθε φορά και πώς μπορεί να εφαρμοστούν Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σημειώσω ένα πρόβλημα το οποίο θα έλεγα θεωρώ θεμελιώδες. Μιλάμε σήμερα για τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της διεθνούς διακυβέρνησης, της σφαιρικής διακυβέρνησης. Οι μηχανισμοί αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι. Βασίζονται στην κυριαρχία την εθνική και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικό μέλος σε ένα πολύ μικρό αριθμό οργανώσεων, σαν παράδειγμα ΠΟΕ, ε, η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, το Κόντεξ Αλιμεντάριος και κάποιες διεθνείς συμβάσεις. Σε κάποιους άλλους διεθνείς θεσμούς, πολύ σημαντικούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ε, σαν ένωση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι άλλο από ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να προσπαθήσουν να έχουν μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ τους και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κληρονομιά. Πρέπει να έχουμε μια εικόνα η οποία να είναι συμβατή με το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει τον ρόλο της και στους διεθνείς οργανισμούς η Ευρωζώνη δεν έχει ας πούμε καμία παρουσία στο IMF, στο ΔΝΤ. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως αυτή η πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και η κυρία Γκόμες, δεν υπάρχει συνήθως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μα τι λέει το άρθρο 13 και το 14 της συνθήκης, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επηρεαστούν και στις, στον τομέα της, του Συμβουλίου Ασφαλείας και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτό. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε πράγματι να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, τις κοινωνικές επιλογές και τις πολιτικές επιλογές, τις οποίες έχουμε αναπτύξει νομοθετικά και σε εθνικά κοινοβούλια και σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ελκυστικότητά μας σε διεθνές επίπεδο, απαιτείται μία φωνή, μία ευρωπαϊκή φωνή και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στον Διεθνή Ναυτικό Οργανισμό. Και η πραγματικότητα είναι ότι σε πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας απλός παρατηρητής μαζί με την κοινωνία των πολιτών και της ΜΚΟ. Πρέπει να αλλάξουν αυτά και νομίζω ότι οι βουλευτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πολλά χάνουμε, ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και να προασπιστούν οι αξίες μας. Μάλιστα. Δεν θα κατάφερνα να καταλήξω σε καλύτερα συμπεράσματα εγώ. Νομίζω ήταν συναρπαστική αυτή η συνεδρία και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μαρτίνες για να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ της συζήτησης. You

Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην τελευταία συνεδρία, στο τελευταίο τμήμα της ε, διάσκεψής μας και παρακολουθώντας τη συζήτηση δεν ε, μπορώ να μην ενδώσω στον πειρασμό και να κάνω και εγώ μερικά σχόλια. Στο τέλος όμως συνεδρίαση θα κρατηθώ μέχρι τότε γιατί έχουμε αρκετά πλήρες πρόγραμμα. Περνάμε επαναλαμβάνω στο τελευταίο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας. Θα μάθουμε πολλά για τις διάφορες οργανώσεις, τα δίκτυα, τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν μεταξύ των κοινοβουλευτικών και που μερικές φορές θα ε, γνωρούμε ακόμη και εμείς. Ακόμη και εμείς που παρακολουθούμε την ε, λειτουργία των δομών και των πρωτοβουλειών της κοινωνίας των πολιτών δεν τα γνωρίζουμε όλα. Πάντως ε, αναζητούνται μορφές συμμετοχής που ίσως μας ικανοποιήσουν περισσότερο από τις υπάρχουσες, ε, τις καθιερωμένες από το κράτος δικαίου εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Στο πάνελ μας έχουμε πολύ έγκριτους ομιλητές για παράδειγμα, έχουμε πρώτη ομιλήτρια την κυρία Σιλβάνα Κοχμερίν, την αγαπητή φίλη που είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για αρκετά χρόνια ήταν και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα εγώ είχα τη μεγάλη χαρά να συμμετέχω μαζί της στις εργασίες του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι και από του τους προτεργάτες μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Φόρουμ των Γυναικών Βουλευτών. Εγώ πραγματικά ε, άσκησα όλη μου την επιρροή και ό,τι πίεση μπορούσα, ώστε και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει την πρώτη μεγάλη τέτοια συνέλευση αυτού του Παγκόσμιου Φόρουμ Γυναικών στα Κοινοβούλια, που συγκέντρωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο πάνω από 500 μέλη. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν θα σας ακούσουμε Σιλβάνα. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Αρνό Λερουά, που είναι μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ε, είμαστε σχεδόν συμπατριώτες θα έλεγα, γιατί ε, εκλέγεται από τους Γάλλους ε, της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Είχαμε βρεθεί και σε προεκλογική εκστρατεία. Ο κύριος Λερουά είναι γραμματέας της Επιτροπής Αιφόρου Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος του Globe Europe, δηλαδή της οργάνωσης ε, που είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Νομοθετών που ασχολείται με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αηφόρο ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Αλέντε Τέσ, που είναι μέλος της Βουλής των Βρυξελών και πρώην πρόεδρος της γνωστής ε, οργάνωσης Κοινοβουλευτική για Παγκόσμια Δράση. Εξακολουθεί μάλιστα να είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο δίκτυο αυτό ο κύριος Αλέντε Τέξ. Και τελευταίος μας ομιλητής θα είναι ο Γιώ Λάινεν, Ευρωβουλευτής με μακροσκελές βιογραφικό, ετέλεσε πρόεδρος πολλών επιτροπών, πολύ σημαντικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι συμπρόεδρος της εκστρατείας υπέρ μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους καλεσμένους μας ε, για να μας παρουσιάσουν τα δίκτυα και τους οργανισμούς τους και θα τους θέρμα παρακαλέσω να είναι σύντομοι γιατί όπως έχετε καταλάβει στις 5.30 πρέπει να εκενώσουμε την αίθουσα. Άλλωστε μερικοί καλεσμένοι μας πρέπει να φύγουν ε, ακόμη πιο νωρίς, στις 5 και 4. Κρίνετε λοιπόν ε, μόνοι σας πόσο χρόνο θα αφιερώσετε στις ομιλίες σας. Σιλβάνα, έχεις πρώτη το λόγο. Σε ακούμε. Uh, Σας ευχαριστώ όλους που μας καλωσορίσατε εδώ. Θα ήθελα να ομιλήσω για το Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Κοινοβουλευτικών. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μίγκελ. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη που έδωσε στο φόρουμ αυτό από την πρώτη στιγμή ήσουν παρόν σε όλες τις διασκέψεις μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την IBU υπάρχουν 9.000 γυναίκες κοινοβουλευτικοί, ο αριθμός είναι πάρα πολύ χαμηλός. Αν δει τις στατιστικές από κοντά δεν είναι ούτε καν το 20% του πληθυσμού των κοινοβουλευτικών στον κόσμο. Και αυτό είναι μια τρομερή αντίφαση σε σχέση με τον πληθυσμό τον οποίο εκπροσωπούν οι βουλευτές αυτές, οι γυναίκες. Βλέποντας λοιπόν τα υπάρχοντα δίκτυα για τις γυναίκες και βλέποντας τι άλλα φόρα υπάρχουν για διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα πολιτικής, πέρα από τα θέματα των δύο τα αυστηρά των σχέσεων κτλ. και αναφέρομαι εδώ στη συνεργασία όλων των γυναικών βουλευτών και όχι μόνο αυτών που συμμετέχουν σε αρμόδιες επιτροπές γυναικών, ήταν καλό να δημιουργηθεί ένα φόρουμ, υπήρχε ενδιαφέρον ανάμεσα στις γυναίκες κοινοβουλευτικούς να συναντώνται και να συζητούν. Αυτό το είδαμε και στο τέλος του Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, όταν κάναμε την πρώτη μας διάσκεψη η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική. Άνω των 500 συμμετεχουσών από 106 χώρες. Φαντάζεστε τον πολιτιστικό πλούτο, τον πλούτο των συζητήσεων, την ευρύτητα των αντιλήψεων. υπήρξε πράγματι μία πλήρης ανάμιξη και η μία γυναίκα ονόμαζε την άλλη αδελφή και υπήρξε μία εξαιρετική και συγκινητική ατμόσφαιρα. Ήταν πράγματι μία πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Και Υπήρχαν βέβαια γυναίκες βουλευτές από όλες ε, τις ε, πολιτικές ιδεολογίες, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είχαν εκλεγεί άμεσα, υπήρχαν ακόμα και εκπρόσωποι από τη Σαουδαραβική Σούρα, υπήρχαν εκπρόσωποι από χώρες τις οποίες έγιναν πολύ πρόσφατα ελεύθερες εκλογές, υπήρξαν εκπρόσωποι από ε, παλαιές δημοκρατίες, και αυτό το οποίο είχε πει η κυρία Μισελ Μπασλέ, η τέος πρόεδρος, η μην πρόεδρος της Χιλής και πάλι και τέος ο πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών. Είχε πει ότι όταν γίνουν πολλές οι γυναίκες ηγέτιδες στον κόσμο τότε θα αλλάξουν και οι κοινωνίες. Αυτό λειτουργήσε σαν φόρουμ λοιπόν, δεν σταθήκαμε αποκλειστικά στα θέματα των διαφορών των φύλων, αλλά προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τις απόψεις των γυναικών. Δεν αποκλείστηκαν οι άνδρες φυσικά, υπήρξαν και αρκετοί ομιλητές άνδρες, κάποιοι από εσά ήσασταν παρόντες στη διάσκεψη τον Νοέμβριο. Αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα σε, τακτία, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα υπάρχουν περιφερειακές διασκέψεις, θα υπάρχουν μελέτες που συμπληρώνουν τις εξαιρετικές εργασίες της IBU στα θέματα των φύλων. Είναι μια προστιθέμενη αξία, αν θέλετε, η οποία αφορά το σύνολο των γυναικών που εκλέγονται στον κόσμο. έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η μειονότητα η κοινοβουλευτική και να φτάσουμε τουλάχιστον στο 50%. Ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι σας ενημέρωσα για αυτό που έπρεπε. Σας ευχαριστούμε κυρία Κοχμερίν και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την σύνεση που και την οικονομία στον χρόνο. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Λερουά για να μας παρουσιάσει την Παγκόσμια Οργάνωση Νομοθετών στην οποία συμμετέχει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση θα σας παρουσιάσω το έργο του Globe και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή για την παρουσίαση. Θα ήθελα να, επαναφερθώ σε, να, επανέλθω σε κάτι που είπε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της Ελλάδας. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της επικοινωνίας και στην ορολογία που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε το πολιτικό μας μήνυμα. Στη Γαλλία πρόσφατα εγκρίναμε ένα ψήφισμα για να προωθήσουμε την διακοινοβουλευτική συνεργασία στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας και μερικές φορές αισθανόμαστε μόνοι μας, απομονωμένοι σε αυτή τη, αυτή μάχη που δίνουμε. Βέβαια, επίκυνται ευρωεκλογέ ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να τολμήσουμε να πούμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε κάποιες μεθόδους συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και μάλιστα ξεκίνησα τη σαρδιδρομία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στον πολιτικό ρυθμό μεταξύ Εθνικού, Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς όταν αναλαμβάνουμε μια νομοθετική πρόταση, ε, ήδη τη λαμβάνουμε σε μεταγενέστερο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας και μερικές φορές κατόπιν εορτής. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ρυθμούς μας, αλλιώς ε, η... θα οδηγήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, σε μια πιο θετική νότα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Νομοθετών ανταποκρίνεται σε μια πραγματική νέα ανάγκη. Η δράση της Globe επικεντρώνεται στην ε, προάσπιση της ε, βιοπικιλότητας, ε, στην προστασία του κλίματος και των δασών. Είμαστε πάνω από 100 χώρες που συμμετέχουμε σε αυτή την Παγκόσμια Οργάνωση Νομοθετών, εκπρόσωποι της, των Άνω και βουλών. Για παράδειγμα, έχουμε και την Globe France που ξεκίνησε στον Ιούνιο του 2012 κατά την έναρξη της θητείας και προσπαθούμε να εγκύπτουμε σε, αυτά τα οικολογικά θέματα με διακομματικό χαρακτήρα και με τέτοια προσέγγιση. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος ε, του Τμήματος Ευρώπης. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα ειδικό τμήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούμε να γίνουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, ένα φόρουμ για να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι μια φράση που την ακούμε πολύ συχνά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν αυτές τις πρακτικές να τις ε, αξιοποιήσουμε και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγαμε στην Κίνα, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ε, της ε, κυβέρνησης για να παρουσιάσουμε τις φιλοδοξίες της Globe. Συμμετείχε μάλιστα και ο Τζον Πρέσκοτ στην αντιπροσωπεία μας. Και φυσικά παρουσιάσαμε και κάποιες εθνικές εμπειρίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψή μας στην Κίνα. Γιατί ενώ εμείς ε, ασχολούμαστε με το backloading του, σύστημα, του συστήματος εμπορίας εκπομπών, οι Κινέζοι μας εξήγησαν ε, το δικό τους μηχανισμό και τα διδάγματα που άντλησαν από τα δικά μας λάθη και τα προβλήματα ελέγχου που αντιμετωπίσαμε εμείς στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, συζήτησης μεταξύ των κοινοβουλίων διεθνώς. Τώρα, υπάρχει αυτή η έννοια του δημόσιου αγαθού, του κοινού αγαθού. Είναι κάτι που ξεπερνά τις κομματικές ή υπερβολικά ιδεολογικές ή συζητήσεις. Το κλίμα είναι ένα κοινό αγαθό. Το 2015 η Γαλλία θα φιλοξενήσει την ΚΟΠ και ήδη ε, προετοιμάζουμε το έδαφος για να αποφύγουμε την αποτυχία. Και νομίζω ότι εκεί η κοινοβουλευτική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Όλε αυτέ οι διαπραγματεύσει είναι αμυγό δια, διακυβερνητικές. Πήγα στα, στο Κατάρ, στη Νότια Αφρική το 2002, στα πλαίσια τη ΚΟΠ και εκεί διαπιστώνουμε ότι οι συζητήσει είναι υπερβολικά τεχνικέ. Δεν γίνονται καθόλου πολιτικέ συζητήσει ε, για τις επιπτώσεις όλων αυτών των συμφωνιών στην καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς ως βουλευτές έχουμε αυτό το καθήκον και αυτή την ευθύνη να επισημάνουμε αυτές τις ανησυχίες. Είχαμε ένα-δύο μήνες σχεδόν πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων και καταιγίδων. Οπότε το θέμα του, της μεταφοράς του πολιτικού μηνύματος είναι πολύ σημαντικό. Εγώ κατάγομαι από τη Ζηρόντα. Χάσαμε 5-6 μέτρα ακτής μέσα σε μία νύχτα σε πολλές περιπτώσεις και μόνο σε μία περιοχή της Γαλλίας. Ενώ οι καταιγίδε ε, παρατάθηκαν για δύο μήνες ολόκληρους. Δυστυχώς ε, έχουν καταστραφεί όχι μόνο θύνες στις ακτές, αλλά μερικές φορές ε, φτάνουν μέχρι τους κήπους και τα σπίτια τα κύματα της θάλασσας εξαιτίας των ακραίων αυτών καιρικών φαινομένων που είχαμε. Ένα άλλο καινούριο στοιχείο, μια νέα καινοτομία, είναι ότι οι σοσιαλιστές που ήταν κάπως διστακτικοί αυτή την, σε αυτό το θέμα, χρειάστηκε να έχουμε έντονες πιέσεις από την κοινωνία των πολιτών για να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Και νομίζω ότι ως ε, βουλευτές έχουμε αυτό το καθήκον ε, να μεταφέρουμε τους φόβους και τις ανησυχίες των ε, πολιτών για τέτοια θέματα και να τις μεταφέρουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Globe είναι μια σχετικά νεοσύστατη οργάνωση. Θα οργανώσει μάλιστα και ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ στο περιθώριο της COP του 2015 και μάλιστα σας προσκαλούμε εκεί. Είχαμε 400 ε, βουλευτές στην αντίστοιχη πρωτοβουλία που κάναμε στο Ρίο, στην προηγούμενη COP και σας καλούμε το Μάρτιο στη συνδιάσκεψη COP που θα γίνει στο Παρίσι το 2015, το Μάρτιο του 2015. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δεστέξ που είναι μέλος του Κοινοβουλίου των Βρυξελών και πρώην πρόεδρος το, του κινήματος ε, κοινοβουλευτική για παγκόσμια δράση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αν δεν τα καταφέρετε εσείς, θα φροντίσω εγώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολύ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι που θα σας παρουσιάσω τους Parliamentarians for Global Action. Είναι μια ενιαία ένωση δραστήρια σε 139 κοινοβούλια στον κόσμο με πάνω από χίλια μέλη βουλευτές. Μια οργάνωση δραστήρια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Είναι μια παλαιά οργάνωση. Ιστορικά δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και για την υπογραφή της συνθήκης εναντίον των πυρηνικών αλλά είμαστε παρόντες και σε άλλους τομείς σήμερα και οι δράσεις μας συνδέονται με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει ένα μορατόριο για την θανατική ποινή στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2014. Πώς το κάνουμε αυτό. Στοχεύουμε ορισμένες χώρες. Φέτος στη Τζαμάικα, το Σουρινάμ, την Κάνα, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνα. Οι χώρες αυτές μέχρι τώρα δεν έχουν υπερψηφίσει το μορατόριο και έρχονται ε, με μια ξεκάθαρη θέση των κυβερνήσεών τους που εμπνέονται από τα κοινοβούλια τους και θα υποχρεωθούν να ψηφιστούν ε, υπέρ αυτού του μορατόριου. Στην περίπτωση της Σενεγάλης, οι χώρες αυτές λέγουν ότι είναι κατά της θανατικής ποινής, αλλά ποτέ δεν έχουν υπερψηφίσει το μορατόριο με επίσημα. Προσπαθούμε λοιπόν έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να, είναι, να έχουν τις θέσεις συμβατές με τις θέσεις που έχουν και σε εσωτερικό επίπεδο. Λοιπόν, οι Parliamentarians for Global Action υποστήριξαν επίσης την προεκλογική εκστρατεία για την επικύρωση της συνθήκης της Ρώμης και της διεθνούς υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 122 χώρες αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στη συνθήκη της Ρώμης και επί 15 χρόνια εμείς βοηθήσαμε στην επικύρωση από 76 χώρες. Πώς ακριβώς εργαζόμεθα. Σήμερα φαίνεται σαφές το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να υποστηρίζεται από μια πλειοψηφία χωρών. Αλλά αυτό δεν ήταν γεγονός πριν 15-20 χρόνια. Σαν παράδειγμα ο Πορτογάλος φίλος που είναι εδώ, ο κ. Μαγκαλάες, είχε οργανώσει στη Λισαβόνα μια πρώτη συνάντηση των Πορτογαλόφωνων χωρών Εκτός από την Πορτογαλία καμία χώρα δεν είχε υπογράψει. Τότε είχαν έρθει όμως οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης στη Βραζιλία, συμφώνησαν στη Λισαβόνα και γύρισαν στη Βραζιλία με μια συμφωνία επικύρωσης. Και έτσι η Βραζιλία επικύρωσε τη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού. Αυτή τη στιγμή το έκανε η Βραζιλία, ήταν πάρα πολύ εύκολο να πείσει κανείς και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής να το κάνουν. Εργαστήκαμε επί μακρόν και για τη Σιλή η Χιλή ήταν πολύ διστακτική λόγω ακριβώς του ιστορικού προηγουμένου του Πινοτσέτ. Εμείς βοηθήσαμε με βουλευτές από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Αργεντινή. Μέσω αυτών των συναδέλφων τους πείσαμε τους χιλιανούς να επικυρώσουν. Ενθυμίστε ότι οι δύο πρώτες ήπειροι ήταν η Ευρώπη βέβαια και μετά η Λατινική Αμερική. Η Ασία είχε μείνει πάρα πολύ πίσω, την έχουμε ξεχάσει σήμερα <coughs> Είχαμε μια συνάντηση στην Ιαπωνία, η ομάδα που δημιουργήθηκε η Εθνική έπεισε την κυβέρνησή της και αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία επικύρωσε, αυτό ξεμπλόκαρε αν θέλετε τη διαδικασία επικύρωσης και για τις άλλες χώρες. Επίσης συχνά σας δίνω αυτά τα παραδείγματα για να σας δείξω ότι είμαστε συγκεκριμένοι και πρακτικοί με συγκεκριμένη δράση και με αποτελέσματα αποδείξιμα. Βλέπουμε ότι μία ολόκληρη σειρά μικρών χωρών δεν είχαν επικυρώσει. Οι Κομόρες, σαν παράδειγμα. Οι Κομόρες δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά πήραμε ένα βουλευτή που συμφωνούσε, γράψαμε τον νόμο για αυτόν, κατέθεσε τον νόμο στο Κοινοβούλιο, δεν υπήρχαν αντιρρήσεις και έτσι και οι Κομόρες επικύρωσαν. Το κάναμε με πολλές μικρές χώρες. <coughs> και έτσι ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 επικυρώσεων. Ε, πάνω από, τα, από τις μισές χώρες δηλαδή έχουν επικυρώσει πλέον τη συνθήκη της Ρώμης. Για να τελειώνω με το διεθνές ποινικό. Ε, η πρόκληση είναι η Αφρική. Ξέρετε ότι με... <coughs> όταν απευθύνθησαν κατηγορίες εναντίον του Μπασίρ, του Σουδάν και του Κενιάτα της Νιγηρίας, απειλείται ουσιαστικά η ύπαρξη του δικαστηρίου στην Αφρική. Εδώ και ένα μήνα η Αφρικανική Ένωση πήρε ένα ψήφισμα, έβγαλε ένα ψήφισμα αρνούμενη συνεργασία με το δικαστήριο. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Γιατί αν χάσουμε την υποστήριξη της Αφρικής, τότε χάνουμε τον καθολικό χαρακτήρα της συνθήκης της Ρώμης και του δικαστηρίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντισταθμίσουμε την επιρροή των κρατών μελών, προσπαθώντας να πείσουμε τους Ευρωπαίους, τους Αφρικανούς βουλευτές, 500 περίπου, ε, να εκφράσουν αντίθετη άποψη από την επίσημη της χώρας τους. Σε πολλές χώρες δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνεις. Μιλάμε για ισχυρά προεδρικά καθεστώτα, τα κοινοβούλια δεν έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε μέσω των κοινοβουλίων να υποδείξουμε στους Αφρικανούς έναν άλλο δρόμο από το ψήφισμα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που είναι αντίθετη με το διεθνές ποινικό. Είμαστε επίσης ε, δραστήριοι και για την σύμβαση για το εμπόριο όπλων που επικυρώθηκε στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε επικυρώσεις από πολλές χώρες την ψήφιση ενός εθνικού νόμου και την εφαρμογή του νόμου. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ανησυχούμε πάρα πολύ για το τι συμβαίνει εκεί σήμερα. Ξέρετε ότι για πολλούς μήνες στρατεύματα πολλές φορές από γειτονικέ χώρες σκότωναν χριστιανούς. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Οι χριστιανοί σκοτώνουν μουσουλμάνους, συμβαίνουν εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, εκαθαρίσεις φυλετικές και κάποιοι μιλούν ήδη και για γενοκτονίες. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να σας προσκαλέσω να πιέσετε έτσι ώστε το ψήφισμα που, βγάλατε, που έβγαλε μάλλον το Συμβούλιο, το, το Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και που επιτρέπει τη χρήση ένοπλης βίας να επιτρέψει σε περισσότερες χώρες να είναι παρούσες στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Γαλλία είναι εκεί παρούσα, είναι σχετικά μόνη της, στηρίζεται επιμελητιακά από το Βέλγιο, τη Σουηδία και την Εστονία, αλλά νομίζω ότι αν πράγματι εμείς στην Κεντρική Αφρική ζήσουμε αυτό το οποίο είχαμε ζήσει στην Ρουάντα πριν πολλά χρόνια, θα είναι μια τεράστια αποτυχία για τη διεθνή κοινότητα και σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε όλοι τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας έτσι ώστε να αποφύγουμε μια τέτοια πιθανή γενοκτονία. Σας ευχαριστώ αλλά θα τελειώσουμε το πάνελ με την παρέμβαση του κυρίου Λάινεν ο οποίος στα πλαίσια και των εργασιών του με τα Ηνωμένα Έθνη δεν ακούω και δεν ξεχνώ ότι ήταν φυσικά και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων όπως επίσης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ καλός γνώστης και έχει προωθήσει στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες οι οποίες ορίζουν την καθημερινότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yeah, Ευχαριστώ πολύ Μικέλ για την ευκαιρία που μου προσέφερες ε, να κάνουμε εκστρατεία με την έννοια ε, να υπάρξει ένα είδος κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχω σε ε, διεθνείς οργανισμούς, είμαι Υπήρξα και εγώ μέλος της κοινοβουλευτικής οργάνωσης Global Action και ε, συμμετείχα επίσης και στις προσπάθειες για να υπάρξει ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Είπαμε σήμερα ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση χρειάζεται το δημοκρατικό έλεγχο. Από πάρα πολλά μέρη του κόσμου υψώνεται, γύρεται το αίτημα να υπάρχει ε, κοινοβουλευτική συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη. Από το 2007 συνήλθαν πολλά άτομα ε, και οργανισμοί έτσι ώστε να υπάρξει κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αποκινούμε άλλους ε, με τον Αντώνη Βιτζιλάντε παραδείγματος χάρη ε, επιδώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη υπογραφές από 1.500 βουλευτές αλλά και από άλλους από <clears throat> κατόχους βραβείου Νόμπελ και άλλους αξιωματούχους που λένε ότι παράλληλα με τις κυβερνήσεις χρειαζόμαστε και τα κοινοβούλια. Ακούσαμε λοιπόν ότι η IPU εδώ και κάποια χρόνια έχει το καθεστώς του παρατηρητή. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόοδο και ε, όσοι εργάστηκαν γι' αυτό πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Τα κοινοβούλια εδώ και 60 χρόνια ε, έχουν συμβάλει στην ύπαρξη των ΗΕ και παρίστανται στις εργασίες των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως εκεί είμαστε παρατηρητές και εγώ πιστεύω κοινοβούλια που έχουν εκλεγεί από τους πολίτες ποτέ δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένα να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όπως η Greenpeace, η Amnesty International ή άλλες ΜΚΟ. Ε, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών και με τη διάδοση της παγκοσμιοποίησης των προβλημάτων αλλά ε, και ε, της ε, μεγαλύτερης επίδρασης των αποφάσεων χρειαζόμαστε το δημοκρατικό έλεγχο. Η Γενική Συνέλευση είναι με βάση το άρθρο 10 το βασικότερο όργανο των Ηνωμένων Εθνών, όμως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν και άλλα όργανα με βάση το άρθρο 22 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι λοιπόν καθόλου δύσκολο να λάβει κανείς την απόφαση ότι θα υπάρχει και ένα παράλληλο όργανο μέσα σε αυτό το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, να υπάρχει δηλαδή μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που γύρεται το αίτημα αυτό, ε, το στηρίζουν ε, πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα θέσψε και σχετικό ψήφισμα στην Ολομέλεια. Το ίδιο ισχύει και για, το, για την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Αφρικανικό, το Λατινικό Κοινοβούλιο έπραξαν αυτό. Ε, κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής, όλοι αυτοί ετάχθησαν υπέρ αυτού του αιτήματο. Και αν δει κανεί ε, με προσοχή την κατάσταση, νομίζω αυτό το βήμα που έκανε η IPU ήταν μια θαυμάσια αρχή που πρέπει να την υποστηρίξουμε. Δεν μπορεί βέβαια να είναι και το τέλος. Το επόμενο βήμα πρέπει να ακολουθήσει και έτσι είτε η IPU θα γίνει αυτό το όργανο, βέβαια στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ε, μεταλλαχτεί από Ένωση Κοινοβουλίων σε Ένωση των Ηνωμένων, ε, σε όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, δύσκολο βέβαια. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε παρόλα αυτά θα πρέπει κανείς να έχει το όραμα ενός οργάνου των Ηνωμένων Εθνών που θα αποτελείται από εκπροσώπους ε, κοινοβουλίων όλου του κόσμου. Αυτά ε, με βάση το άρθρο 22 των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν θα επηρεαστεί κανένα άλλο όργανο των ΗΕ. Θα συνεχίσει να υπάρχει η ε, Γενική Συνέλευση και ο Γενικός Γραμματέας. Αυτή λοιπόν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα, ακριβώς όπως υπάρχει και στο ε, Συμβουλίο της Ευρώπης και όπως ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα πλεονεκτήματα βεβαίως είναι σαφή. Εάν οι βουλευτές του κόσμου συνήρχονται, τότε θα συζητούντο τελείως διαφορετικά τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή, κάτω από διπλωματικό, με κοινοβουλευτικό και όχι διπλωματικό πρίσμα. Αυτοί οι βουλευτές θα μπορούσαν να υποβάλουν επερωτήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και προς άλλους ε, ε, αξιωματούχους των ΗΕ και με τον τρόπο αυτό να ρίξουν φως στα προβλήματα του κόσμου θα μπορούσαν να οργανώσουν ακροάσεις, να συντάξουν συστάσεις. Επίσης ε, θα μπορούσαν λίγο σε πιο προχωρημένο στάδιο να ελέγχουν ε, πώς ακριβώς ε, χορηγούνται τα κονδύλια των Ηνωμένων Εθνών. Με λίγα λόγια δηλαδή υπάρχουν πολύ προχωρημένες ιδέες για το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά μια τέτοια κοινοβουλευτική συνέλευση δεν μπορεί να είναι το κογκρέσο της Κίνας με 3-4 χιλιάδες βουλευτές. Ε, θα πρέπει να είναι ένα όργανο από 700 μέχρι 900 βουλευτές. Κάθε χώρα θα έστελνε δύο βουλευτές για να συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Τίθεται βέβαια το εξής ερώτημα. Υπάρχουν χώρες όπου δεν έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα, έχουν δικτατορία. Και τι θα γίνει με αυτές, θα συμμετέχουν. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι και μέλος ε, της ΑΚΕ, και βλέπω ότι εκεί υπάρχουν χώρες οι οποίοι δεν έχουν ρετούς εκπροσώπους. Και παρόλα αυτά οι χώρες αυτές εκπροσωπούνται στην ΑΚΕ με εκπροσώπους των χωρών τους, άρα δηλαδή ένα τέτοιο όργανο θα προήγαγε τον εκδημοκρατισμό και τον κοινοβουλευτισμό ανά τον κόσμο. Μόλις πριν από λίγο έγινε λόγος για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τη δεκαετία του 70 και του 80 αυτό ήταν ε, η απόλυτη ουτοπία, έτσι αντιμετωπίζεται, και σε λίγα όμως μόνο χρόνια ε, συνετάχθησαν τα, το, συνετάχθη το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικατικού Δικαστηρίου, γιατί όχι και για την IPU και εκεί μπορεί να συμβεί το ίδιο. Εύχομαι λοιπόν με αυτή τη σημερινή μας συνάντηση και πολλές άλλες που θα ακολουθήσουν ε, στο τέλος της δεκαετίας να έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο έτσι ώστε ή να γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών ή να κάνουμε ξεχωριστά αυτό το όργανο που οραματιζόμαστε και στο τέλος του αιώνα να συνδυάσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση με την παγκόσμια δημοκρατία που νομίζω είναι κάτι που θα μας ενώσει όλους μας. Θερμά ευχαριστώ, Γιώ. Θα περάσουμε τώρα στο γύρο των ομιλητών. Δεν είναι πολύ, γιατί περισσότερο έγινε αυτή η διάλεξη για να συγκεντρώσουμε κάποιες, κάποιες πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες τις ακούσαμε χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να τις αφομοιώσουμε. Άλλωστε μεταξύ έφυγαν και κάποιοι συνάδελφοι, οπότε λίγοι είναι αυτοί που ζήτησαν το λόγο. Πρώτα θα μιλήσει η κυρία Γκαμπριέλα Κρέτσου, γερουσιάστρια από τη Ρουμανία και πρώην ε, Ευρωβουλευτής και πολύ αγαπητή φίλη. Γκάμπι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ θερμά, Μιγγέλ.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 ε, και η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό ε, συναντιόμαστε σε διεθνές επίπεδο, σε συναντήσεις. Παρόλα αυτά όμως ε, εξακολουθούμε να περιοριζόμαστε σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω δηλαδή ότι μια κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ε, θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική εφόσον δεν ε, μετεξελίσσονται τα πολιτικά κόμματα. Και όσο δηλαδή δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε πολιτική. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας μπλοκάρει ένα είδος ε, πολιτικής ε, συζήτησης, ε, τυποποιημένης πολιτικής συζήτησης. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση των γυναικών που έλαβε χώρα τον Οκτώβρη και όπου συμμετείχα, όσοι πραγματικά έδωσαν τον τόνο προήρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Εγώ υποστηρίζω στεναρά τον κοινοβουλευτισμό, αλλά δεν νομίζω ότι η κατάσταση θα αλλάξει όσο αυτά τα φόρα εξακολουθούν να υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως ε, και θα αποκτήσουμε περισσότερες ε, σχέσεις με συναντέλφους ανά τον κόσμο. Αλλά ειλικρινά διαρωτώμε κατά πόσο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή. Γιατί σε τελική ανάλυση το πρόβλημα εμφανίζεται λίγο πριν από μία ε, δεσμευτική πολιτική ε, απόφαση. Τα εθνικά κοινοβούλια τελικά είναι υπό την καθοδήγηση των κυβερνήσεων. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση χρειαζόμαστε δημοκρατικούς θεσμούς στο κατώτατο επίπεδο και μετά πρέπει ε, να ανέβουμε προς τα πάνω. Γιατί αλλιώς θα φτιάξουμε μόνο οργανώσεις ε, οι οποίες θα ευνοούν παράνομες αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρέτσου. Ο τώρα στον συνάδελφο Κάλβιντς από τη Λετωνία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές και κυρίως ε, τη Σιλβάνα Κοχμερίν που μίλησε για το ρόλο των γυναικών. Η Λετωνία είχε γυναίκα πρόεδρο. Η πρόεδρος της Βουλής της Λετωνίας ε, είναι γυναίκα και επίσης μόλις εκλέξαμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό. Οπότε ίσως ένας από τους λόγους που ε, επέτυχε οικονομικά η Λετωνία είναι ότι αναγνωρίζει όλο και περισσότερο το ρόλο των γυναικών ε, στην χώρα. Κάτι που δεν αναφέρθηκε παρκώς είναι το θέμα των νέων. Η νεολαία. Μία από τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες ε, διαδηλώσεις της Βορείου ξεκίνησαν από άνεργους νέους, από νέους κάτω των 30 ετών. Και ενώ σε πολλά μέρη της Ευρώπης έχουμε πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού, σε πολλά μέρη του κόσμου το πρόβλημα είναι αντίστροφο. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να εμπλέξουμε περισσότερο τους νέους στην όλη διαδικασία. Γιατί ναι, μεν, όταν βλέπουμε τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, διαπιστώνουμε ότι η χαμηλή αυτή συμμετοχή αγγίζει και τους νέους, ε, ίσως γιατί ούτε και αυτοί ενδιαφέρονται για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην νεολαία μας, να την εμπλέξουμε και να την προετοιμάσουμε γιατί ό,τι είδους παγκόσμια διακυβέρνηση και να ετοιμάσουμε θα την κληροδοτήσουμε στους νέους και αυτοί θα πρέπει είτε να τη διορθώσουν είτε να την διαχειριστούν και να την ασκήσουν αυτή την παγκόσμια διακυβέρνηση. Ευχαριστώ, δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους του πάνελ για να σχολιάσουν ε, αυτά που μας είπαν οι δύο μιλητές μας και ενδεχομένως ε, να σχολιάσουν και τις ομιλίες που άκουσαν ε, καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Τώρα θα αλλάξουμε τη σειρά των ομιλητών και θα δώσω πρώτα το λόγο στον τελευταίο ομιλητή από το, από το πάνελ μας, τον Γιολάινα δηλαδή. Παρακαλώ όμως να μην μακρηγορήσετε, απαντήστε. Άντε μακρηγορήστε, αλλά μην μακρηγορείτε πολύ τουλάχιστον. Η Γκαμπριέλα έθιξε το πρόβλημα ότι αν τελικά σε ευρωπαϊκό και αργότερα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε βουλευτές ε, αν υπάρχουν βουλευτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, πώ μπορεί αυτό να λειτουργήσει, πώ θα το δεχτεί, δεχτούν ε, οι πολίτες ε, και πώ θα υπάρχει επαφή με, τις, ε, με τα κράτη προέλευση. Τώρα, όσον αφορά τον ενδεχόμενο κοινοβουλευτική συνέλευση των ΗΕ, αυτό θα έχει το πλεονέκτημα ότι οι βουλευτέ δουλεύουν διαφορετικά από του διπλωμάτε. Μιλάνε με μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο άμεσα, διατυπώνουν ιδέες, προτάσεις και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή ε, θα μπορούσαν να ε, διαμορφωθούν και τα διάφορα πολιτικά ρεύματα, συντηρητική, προοδευτική, φιλελεύθερη. Δηλαδή ο κόσμος θα αποκτούσε πολιτικό πρόσωπο με όλα αυτά τα ρεύματα. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυναμική που θα ενδιέφερε και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι σε χώρες όπου δεν υπάρχει δημοκρατία ή είναι ε, σάπιες οι δημοκρατικές δομές, ε, πράγματι ε, πολλοί δεν εμπιστεύονται τους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Στις δημοσκοπήσεις οι διεθνείς οργανισμοί έχουν μερικές φορές μεγαλύτερη αξιοπιστία από ό,τι οι εθνικοί. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλάντε Στέξ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στην συνάδελφα από τη Ρουμανία ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Το θέμα είναι να σκεφτόμαστε παγκοσμίω και να δρούμε τοπικώς. Αυτό όμω δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί κάθε χώρα είναι διαφορετική. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του. Όλοι είμαστε επιπισμένοι ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τη θανατική ποινή, αλλά όταν προσπαθούμε να το εξηγήσουμε ακόμη και σε συναδέλφους από το Κονγκό, γιατί εγώ έχω στενές συνεργασίες με Κονγκολέζους βουλευτές στην Κενσάσα και είναι δύσκολο, γιατί πολλοί από τους βουλευτές του Κονγκό θεωρούν ότι είναι καλή η θανατική ποινή. Δεν συμφωνώ με την κατάργηση. Οπότε και οι βουλευτέ ε, δεν μπορούν να είναι πλήρω αποσυνδεδεμένοι από το σφιγμό και τον παλμό του πληθυσμού τη κοινωνία του. Οπότε σίγουρα πρέπει να δρουν τοπικά και παρά το δικό του όραμα και τη δική του προοπτική θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το σφιγμό και την κρατούσα γνώμη της κοινωνίας του λαού. Αναφέρθηκε το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σχεδόν όλη η Λατινική Αμερική κύρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μόνο κάποιες χώρες της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συμφωνία. Το Σαλβαντόρ, για παράδειγμα, ή η Νικαράγουα. Μικρές μένει χώρες και υπόλοιπε χώρε τη Λατινική Αμερική έχουν ακυρώσει το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Το θέμα είναι αν τοπικά υπάρχουν μεγάλε αντιστάσει, είναι δύσκολο ε, να κατανικηθούν. Δίκιο πάντω έχει και ο συνάδελφο για την νεολαία. Είναι δύσκολο να εμπλέξουμε τους νέους σε όλα αυτά τα θέματα. Ακόμη και στις εθνικές πολιτικές είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία διαπιστώνουμε αυτή την απροθυμία των νέων. Και ίσως η Ροάντα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τόσες πολλές γυναίκες στο κοινοβούλιο της. Εν μέρει όμως αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ένα μεγάλο τμήμα του κοινοβουλίου ε, εκλέγεται από το σύνολο του πληθυσμού, αλλά για ένα μικρό τμήμα ισχύουν ποσοστώσεις. Ποσοστώσεις για τις γυναίκες, για τα πανεπιστήμια, για τους αναπήρους και για τους νέους. Οπότε αυτό αυξάνει τη συμμετοχή των γυναικών στη Βουλή της Ρουάντας. Δεν λέω να κάνουμε το ίδιο, είναι δύσκολο να εμπλέξουμε τους νέους, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Αρνό Λεγουά. Ευχαριστώ, Μίγκελ Εγώ προσπάθησα να πω στην εισαγωγή μου ότι με ενδιαφέρει η η επαφή με την πραγματικότητα. Οι κοινοβουλευτικέ δράσει δεν θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένε από την πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να βρούμε λύσει στα πραγματικά προβλήματα. Και φυσικά να συμφωνήσουμε στη διάγνωση. Γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα, Γιατί υπάρχει αυτή η κρίση στην εκπροσώπηση που ισχύει και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Εγώ βέβαια εκπροσωπώ του Γάλλου που διαμένουν εκτό τη Γαλλία, αλλά είναι επίση φορείς της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά και για απλά θέματα, όπως η έκδοση ταυτότητας, έχουμε προβλήματα γιατί είναι αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην Πορτογαλία και ακόμη υποχρεωμένο να πηγαίνω στην πρεσβεία, στο προξενείο, για την ανανέωση της ταυτότητάς μου. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πολιτική πραγματικότητα που δυστυχώς ε, η πλειοψηφία των πολιτών δεν την αντιλαμβάνεται. Και λαμβάνω ως παράδειγμα την Ιβυρική Χερσόνησο που διανύει χαλεπούς καιρούς. Όταν μιλούμε σήμερα για εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, ενώ ο κόσμος γνωρίζει ότι όλα ε, γίνονται από την Τρόικα χωρίς καμία δημοκρατική νομοποίηση, το συζητήσατε και εδώ, ε, θα πρέπει να κάνουμε ένα έργο διαπαιδαγώγησης ε, για να ξαναπείσουμε τον κόσμο για το, την αξία που έχει ο κοινοβουλευτισμός και για το θέμα των νέων. Ε, και εγώ είμαι στην ομάδα των Ευρωβουλευτών που είναι κάτω των 40, που είναι ελάχιστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δίνουμε μάχη και στη Γαλλία. Προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τώρα το συνταξιοδοτικό μας. Υπάρχει όμως ε, ε σύγκρουση μεταξύ των γενεών. Μεταξύ εκείνων που είναι της παλιάς γενιάς πάνω από 55 και τον ε, της νέας γενιάς στη Γαλλία που δεν είναι εύποροι όπως οι πιο ηλικιωμένοι και έχουν πρόβλημα να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Και είμαστε πολύ μικρή ψηφία στο κοινοβούλιο. Και στην Ισπανία, πήγα στην Ισπανία για το, για το κίνημα των αγανακτισμένων. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθεί και ποια θα είναι η πολιτική διέξοδος. Αλλά ελάχιστη ήταν, ελάχιστες ήταν οι ευκαιρίες για πολιτική διέξοδο, οπότε είναι λογικό να μην επιδιώκουν οι νέοι να εμπλακούν στην πολιτική και να εκλεγούν. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό και αν δεν το φροντίσουμε θα έχουμε δυσκολίες μετά από 10-15 χρόνια. Θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο μας και να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι η νεολαία είναι προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική, μακάρι. Όταν βλέπω στο θέμα της εγγύησης των νέων, βλέπω ότι δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί εμπράκτος αυτό στις διάφορες περιοχές της Γαλλίας, ποιος θα είναι επιλέξιμος για να υποφεληθεί από αυτήν την εγγύηση των νέων. Και υπάρχει και το θέμα της αμεσότητας της δράσης, της ταχύτητας δράσης, γιατί η κατάσταση για την νεολαία είναι κρίσιμη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στις πιο ευάλωτες. Και βλέπουμε και σημαντική μετατόπιση της ισπανικής νεολαίας προς τη Γερμανία, για παράδειγμα μετανάστευση και υπάρχει θέμα ίσως διακρατικών αποζημιώσεων εδώ. Ναι, με να δώσουμε προτεραιότητα στους νέους, αλλά να φροντίσουμε ώστε να αναλάβει νεολαία στα χέρια της το πεπρωμένο της. Γιατί υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού λόγου και της πραγματικής κατάστασης της νεολαίας που δεν θεωρεί ότι εκπροσωπείται δεόντως από τους πολιτικούς. Επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ποια είναι η διάγνωση που κάνουμε για την κατάσταση και πού οφείλεται αυτή η δυσπιστία και η καχυποψία απέναντι στις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις. Ευχαριστώ Αρνό και θα ολοκληρώσουμε αυτό το γύρο των απαντήσεων κατά κάποιο τρόπο των μελών του πάνελ μας με την Σιλβάνα Κοχμερίν και στη συνέχεια θα αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Η Σιλβάνα. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ στο θέμα των νέων. Είναι ένα αιώνιο θέμα, αν θέλετε. Διαπιστώνουμε ότι οι νέοι σήμερα δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι, δεν ασχολούνται με την πολιτική. και το ίδιο έλεγαν και οι γονείς μου για μένα και οι γονείς τους για τους γονείς μου και τα λοιπά. Κάθε νέα γενεά βλέπει με διαφορές ε, τις προηγούμενες και πιστεύει ότι οι νέοι κάθε φορά ίσως να μην είναι απόλυτα αξιόπιστοι και κάτι θα πρέπει να γίνει για αυτούς. Λέγεται επίσης στα γερμανικά περισσότερο ότι οι σημερινές άσχημες ε, εποχές είναι οι καλές εποχές για το μέλλον μας. Εγώ δεν θέλω να σμικρίνω το πρόβλημα, δεν θέλω επίσης να το αποκρύψω, αλλά ιδιαίτερα για το ρόλο των γυναικών στο Global Forum, να πω ότι αυτό το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε είναι να δούμε την πολιτική καριέρα σαν μια προοπτική επιλογή για τις γυναίκες. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει και οι γυναίκες, τα νέα κορίτσια να βλέπουν τους εαυτούς τους σαν πιθανές πολιτικούς, σαν πιθανούς βουλευτές. Και αν δεν το κάνουν αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς η ίδια ιστορία. Σύνεπώς λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κοινοβούλια θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αν είσαι γυναίκα κοινοβουλευτικός, είσαι πρότυπο, είσαι ηγέτη στην κοινωνία και είναι κάτι το αρκετά επαναστατικό να βλέπουν τις γυναίκες οι νεότεροι να ψηφίζουν νόμους και να φροντίζουν για την εξέλιξή τους. Πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να έρθουν σε επαφή με τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό θα αλλάξει τις αντιλήψεις, αυτό θα ανοίξει τις επιλογές για τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον τους και αυτό πρέπει να ξεκινήσει όσο πιο νωρίς γίνεται. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Running Start και η οποία δουλεύει με νέα παιδιά και νέα κορίτσια και αναφέρει από μικρή ηλικία τις ικανότητες που πρέπει να έχουν για να ενδιαφερθούν για την πολιτική. Θα ήθελα και το Global Forum των γυναικών να δουν ακριβώς τι ε, μπορεί να γίνει ως προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα γιατί σε ευρύτερε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. εάν δείτε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, πράγματι είναι παγκοσμιοποιημένες. Τα οικονομικά θέματα, τα οικονομικά, τα χρηματοδοτικά. Θα δείτε ότι ο κόσμος δεν έχει σύνορα πια. Οι κεφάλαια αγορές δεν έχουν σύνορα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν έτσι και αλλιώς και αυτές σύνορα. Οι πολυεθνικές Άκουσα ότι είναι εκατομμύρια ο δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός του Βελγίου μαζί με τις συντάξεις και αν δει κανεί τον κύκλο εργασιών μιας μεγάλης ε, εταιρείας ε, γερμανικής ε, στη Γερμανία της Daimler θα δει ότι ξεπερνάει τα 100 δις και φτάνει τα 115. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Τζο Λάινεν και άλλων έτσι ώστε οι αποφάσεις γύρω από τα θέματα αυτά να μην αφήνονται αποκλειστικά μόνο στους διπλωμάτες και στα μέλη του εκτελεστικού αλλά να ελέγχονται δημοκρατικά. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται σήμερα, αλλά χρειάζεται μία προοπτική, είναι κάτι που πρέπει να συμβεί, θα πρέπει οι βουλευτές να λειτουργήσουν σωστά και σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ Σιλβάνα. Συνάδελφοι, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα πλέον ε, στο τέλος ουσιαστικά της συνάντησής μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η οποία θα εμπνεύσει πολλούς από μας. Κανονικά θα έπρεπε ίσως να τελειώσει με μια ομιλία του κυρίου Καράς και θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω να μου δώσετε τη δυνατότητα κάποιες σκέψεις θέλω να προκαλέσω κάποιες συζητήσεις, αλλά θέλω να συνεισφέρω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι για πολλούς από μας η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών οδηγεί στην ένωση όλων των χώρων του κόσμου και αυτό ταυτίζει τις ε, λαούς του κόσμου με τις κυβερνήσεις του κόσμου έχουμε περάσει σε μια διαστροφή να μιλάμε για διακυβερνητικές οργανώσεις ε, αντί να μιλάμε για διακρατικές οργανώσεις. Μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τους λαούς του κόσμου δεν μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από τους κυβερνήσεις αυτών των λαών, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν και οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των λαών του υπόλοιπου κόσμου. Λοιπόν όλα αυτά στην ουσία ρίχνουν νερό στο μήλο συναδέλφων οι οποίοι μας έδειξαν με τις εμπειρίες τους και με τον ενθουσιασμό τους, ένα θαυμαστό ενθουσιασμό, άξιο θαυμασμού επαναλαμβάνω και αναγνώρισης. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας κατάστασης συζητώντας. Και η συζήτηση μερικές φορές φάνηκε να είναι επανάληψη προηγούμενων συζητήσεων. Είναι σαν το κογκρέσο των Βερσαλιών που έγινε πριν από πολλές δεκαετίες. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρούμε δύο φαινόμενα εδώ. Ως βουλευτές δεν μπορούμε να γνωρούμε τα εξής δύο φαινόμενα. Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό τμήμα των συμπολιτών μας, του εκλογικού σώματος, των λαών και κυρίως των νέων μας, έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη σε αυτό που εμείς εκπροσωπούμε. Γιατί η πλειοψηφία των συμπολιτών μας και κυρίως των νέων πολύ σωστά έχουν την εντύπωση ότι οι περισσότερες αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τα κοινοβούλια αλλά από τις τράπεζες και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση τα κοινοβούλια είναι ε, εργαλεία για την υλοποίηση των πολιτικών που επιβάλλουν αυτές οι τραπεζικές ε, ε, ενώσεις ή τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πώς λοιπόν θα έχουν εμπιστοσύνη σε, στα κοινοβούλια αφού ταυτίζουν τα κοινοβούλια με την πλήρη ανικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε, να επιλύσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι μια διάγνωση, μια διαπίστωση σχεδόν αδιάσυστη γιατί ναι, συζητούμε τα εθνικά κοινοβούλια, νομιμοποίηση και που, σε τι επίπεδο θα πρέπει να έχουμε την νομιμοποίηση. Τις προάλλες άκουσα έναν πολύ σημαντικό στοχαστή από το Βέλγιο που έλεγε πώς τα εθνικά κοινοβούλια είδαν να μειώνονται οι αρμοδιότητες τους γιατί αυξάνονταν οι αρμοδιότητες των περιφερειακών κοινοβουλίων, οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ συρρυκνώνονταν όλο και περισσότερο οι εξουσίε και αρμοδιότητε των Εθνικών Κοινοβουλίων για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Γιατί αυτά τα προβλήματα αναλύονταν και συζητώνταν είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντω ε, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτή η κατάσταση μας οδηγεί στον κρεμό που είναι η άρνηση όλων αυτών των αξιών, η κατάρρευση όλων αυτών των αρχών που στήριζαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μας. Τώρα, ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Κάποιος πολύ εύστοχα επισήμανε ότι η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να εδραιωθεί ως παγκόσμιος παράγοντας, τι να σου πω, στο παγκόσμιο προσκήνιο δεν εδερώσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο παίκτη, τότε θα μείνει έξω από το παιχνίδι. Γιατί άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες θα διαχειριστούν την ειρήνη, την οικονομία ή την κοινωνική πρόοδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη. Αυτό όμως δεν θα το καταφέρει γιατί οι οικονομικές εξουσίες είναι αυτές που, λαμβάνουν τις αποφάσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες δεν έχουν κανένα συμφέρον να καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος ε, παίκτη. Το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη, το, μόνο, το πρώτο που θα κάνει είναι να προσπαθήσει να ανακτήσει αυτό που υπήρχε σε εθνικό επίπεδο και εξαφανίστηκε και καταργήθηκε. Δηλαδή να, να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στις δραστηριότητες αυτών των ε, τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ε, δυνάμεων. Τη διαφάνεια και τον σχετικό έλεγχο ή την υπαγωγή τουλάχιστον αυτών των ε, δυνάμεων σε συγκεκριμένες δημοκρατικές λειτουργίες και κοινωνικές αξίες. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις, οι τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές, που καθοδηγούνται αποκλειστικά και μόνο από το κέρδος και το προσωπικό τους, δικό τους όφελος, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να εγκαθιδρυθεί μία εξουσία που θα αποκαταστήσει τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την υπαγωγή τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές αξίες και δημοκρατικές αξίες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των νέων μας προς τη δημοκρατία και προς την πολιτική και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθιέρωσή της ως παγκόσμιο παίκτη, αν δεν καταφέρουμε πρώτα να ανακτήσουμε την πραγματική νομιμοποίηση και την επιστροφή της, της εξουσίας λήψης αποφάσεων στα κοινοβούλια. Γιατί την έχουμε χάσει αυτή την εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές ευρωεκλογέ σε τρεις-τέσσερις μήνες μόνο. Χθες σε μία συζήτηση με πολλούς ε, συντρόφους, πολλοί ήταν Γερμανοί μάλιστα, έβαλε ένα στίχημα. Έβαλα στίχημα ότι δεν θα καταφέρουμε ούτε 40% συμμετοχή στις ε, ευρωεκλογέ φέτος. Και σε πάνω από 15 χώρες θα έχουμε ποσοστό συμμετοχής κάτω από 30%, δηλαδή 70% αποχή. Και μάλιστα αυτό μια στιγμή που οι βουλευτές, όσοι θα εκλεγούν σε αυτές τις εκλογές, θα έχουν πολύ περισσότερες εξουσίες ε, από οποιοδήποτε κοινοβούλιο προηγουμένως, ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόκληση και σε αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας και δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια οξυδερκή διάγνωση της κατάστασης. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι για παράδειγμα στην πατρίδα μου, στην Ισπανία, κάτι πολύ βασικό, να κλείνουν 7 εργοστάσια της coca ενώ είχαν υπέρογκα κέρδη. Και κλείνουν αυτά τα 7 εργοστάσια γιατί δεν τους συμφέρουν. Και έτσι μένουν 15.000 άτομα χωρίς δουλειά από τη μια μέρα στην άλλη. Μόνο και μόνο επειδή η Coca-Cola αποφάσισε ότι δεν έχει αρκετά κέρδη και προτιμά να μετεγκαταστήσει τα εργοστάσια της, γιατί συμφέρει να τα βάλει αλλού. Φυσικά τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να, να τις καταλάβουν οι συμπολίτε μας, εκτός και αν είναι μέτοχοι οι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola. Πόσοι συμπολίτε μας όμως έχουν τέτοιες θέσεις και αξιώματα. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκλησή μας. Να ανακτήσουμε για τον κοινοβουλευτικό θεσμό, για τη δημοκρατία και την πολιτική, την αξιοπρέπεια που σημαίνει να αποφασίζουμε για τη μοίρα και την πραγματικότητα των συμπολιτών μας. Και θα ολοκληρώσω με μια προσωπική εμπειρία. Είμαι 37 χρόνια βουλευτής, 22 στην Εθνική Βουλή και 15 χρόνια ευρωβουλευτής. Πριν από 35 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, όταν μερικοί ξεκινήσαμε να ξαναφτιάχνουμε τη δημοκρατία στην ε, Ισπανία, εγώ γύριζα στην, στις διάφορες περιφέρειες και περιοχές της Ισπανίας και είπα ποιους θα προτείνω για δημάρχους, ε, για περιφερειάρχες, ε, για βουλευτές και έψαχνα τους καλύτερους και κανένας ποτέ δεν μου είπε όχι. Πάντα μου έλεγαν ότι θα είμαι ικανός και θα τα καταφέρω. Την ίδια εμπειρία την επαναλαμβάνω σήμερα. Πηγαίνω στα ίδια χωριά, στου ίδιου Δήμου και κοινότητε και λέγω στο δάσκαλο, στην, στο γιατρό, στην νοσοκόμο, στον ναυτικό. Λέω, θα ήθελα να είσαι ο υποψήφιό μα ε, στι ευρωεκλογέ. Και μου λένε, καλά τρελάθηκε, έχασε τα μυαλά σου. Εγώ είμαι μέλο του κόμματο, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ υποψήφιο. Άφησε με στην ησυχία μου γιατί θέλεις να αναλάβω εγώ τέτοια καθήκοντα, αφού μια χαρά είμαι, στην ησυχία μου, στο επάγγελμά μου, στο μαγαζί μου. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου οι υποψήφοι δεν είναι πια οι καλύτεροι, γιατί οι καλύτεροι αρνούνται την υποψηφιότητα, αλλά είναι απαράτσι και είναι κομματικά όργανα και κομματικά στελέχη. Και βρίσκουν στην πολιτική μια δραστηριότητα σχετικά αποδοτική και καλά αμοιβόμενοι, αλλά οι καλύτεροι, οι πιο εκλεκτοί των πολιτών μας δεν θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και ένας συμπατριώτης μου που ήταν και βουλευτής μου είπε ότι ένας δικός του συνάδελφος και μάλιστα από τη μετριοπαθή δεξιά της χώρας με υψηλά αξιώματα, ήταν, έφτασε ως και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, πολύ καλός άνθρωπος, τελικά για κομματικούς λόγους δεν ε, έγινε καν βουλευτής, δεν μπήκε στο ψηφοδέλτιο και το ρώτησα, έχεις καμία νοσταλγία? Καμία μου λέει. Για 15 χρόνια είχα μία Mercedes και έβλεπα να γράφουν στους στίχους, κλέφτη, με αυτά που κλέβεις από τον κόσμο αγοράζεις Mercedes. Τώρα έχω την ίδια Mercedes, δεν είμαι πολιτικός, είμαι δικηγόρος, άνοιξα το δικηγορικό μου γραφείο και κανένας δεν λέει ότι έκλεψα. Λέει ο κόσμος, α, αυτός πρέπει να είναι πολύ καλός δικηγόρο, γιατί κατάφερε και αγόρασε Mercedes. Τη Mercedes που για πολλά χρόνια την είχα ω αιτία για στίγμα, για προσβολή και ύβρι, έγινε ουσιαστικά διαφημιστικό εργαλείο. Και προσέλκυε και νέους πελάτες γιατί ο κόσμος σκεφτόταν ότι θα είμαι καλός δικηγόρο. Αυτά λοιπόν στη ζωή μας αγώνα για την ελευθερία έκφρασης και έχουμε πραγματικά το παράδοξο αυτά τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βρίσκονται στα χέρια εκείνων που δεν θέλουν να εδραιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη. και συμβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών εκείνων των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν την πολιτική και προσπαθούν να υπηρετήσουν και τους συμπολίτε τους. Και σε τελική ανάλυση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελάχιστα εξυπηρετούν τη δημοκρατία. Ενώ όλοι πιστεύαμε ανέκαθεν ότι η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν θεμέλιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την προσοχή σας και μακάρι να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις και να συμφωνήσουμε όλοι στην ανάγκη ανάληψης κοινή δράσης για να διασώσουμε και να, τη δημοκρατία, να διαφυλάξουμε την πολιτική και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που είναι πιο σημαντικό από ποτέ και όλος παραδόξως ε, ε, πιο απειλούμενο από ποτέ. Σας ευχαριστώ.